certain uh, groups Uh, good afternoon, everybody. If I could have um, your attention. Καλησπέρα σας. Ε, μπορώ να έχω λίγο την ε, προσοχή σας. Κύριο Ζουβάν, θέλω να ξεκινήσω τη συνεδρίαση. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην πρώτη από τις τρεις συνεδρίες της Επιτροπής μας ε, αυτή την εβδομάδα σήμερα το απόγευμα και αύριο πρωί και απόγευμα. Αύριο θα ψηφίσουμε και όλα για σημαντικέ προτάσει. Θα αρχίσουμε στι 9.45 αύριο το πρωί την ψηφοφορία. Σα το λέω, 9.45. Θα αλλάξω ένα μικρόφωνο, το μικρόφωνο γιατί φαίνομαι καλύτερα στο ίντερνετ αν αλλάξω. Είναι καλύτερη η εικόνα μου. Λοιπόν, αύριο 9.45 ψηφίζουμε. Και αύριο το απόγευμα στις 3 η ώρα μέχρι τις 5 Έχουμε μια σημαντική ακρόαση για πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του διαδικτύου και των πληροφοριών και το σχετικό κανονισμό ή οδηγία, δεν ξέρουμε ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρωτοβουλία για την ασφάλεια του διαδικτύου και των πληροφοριών, πολύ σημαντική. Σα ενημερώνω και γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω όλους όσους μας βλέπουν ε, στο διαδίκτυο. Έχει πάρα πολύ υγρασία ε, σήμερα στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να βγει ο ήλιος πιο μετά. Εδώ έχουμε και παράθυρο άλλωστε και μπορούμε να βλέπουμε έξω, ενώ σε άλλες αίθουσες δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, για τα Για τα τυπικά μας τώρα, ξέρετε ότι βγαίνουμε στο διαδίκτυο ζωντανά. Στείλαμε σε εσά ένα σημείωμα για την πρόσφατη αποστολή μα στη Λιθουανία εν ώψη τη Λιθουανική Προεδρία, με την οποία συζητήσαμε πολλά πράγματα για τη μελλοντική του εργασία στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά και στα ιταλικά και μπορείτε να το βρείτε και στο ιστότοπο, στον ιστότοπό μα μπορείτε να το διαβάσετε. Υπάρχουν επίσης και τα επίσημα πρακτικά της 7ης Μαΐου, της δικής μας συνεδρίασης. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά, θα θεωρούν εγκεκριμένα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αν δεν ακουστούν αντιρρήσεις ή σχόλια. Να περάσουμε τώρα σε ενημέρωση, ε, κάτι το οποίο κάνουμε συνεχώς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Ιρλανδική Προεδρία. Το ξεκινήσαμε πριν από τα Χριστούγεννα για την, πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ε, σε τριμερείς διαλόγους. Ε, Καλώ τους ε, εισηγητές μας να μας ενημερώσουν πού βρισκόμαστε με τις διάφορες προστάσεις. Βερνιό, Ταραμπέλα και Ζουβάν είναι εδώ παρόντες, τους καλωσορίζω. Και εγώ θα σας πω για τη δική μου έκθεση και θα μιλήσω και εκ μέρους της κυρίας Ρόιτοβα. Οπότε ας ακούσουμε μια σύντομη ενημέρωση από τους συναδέλφους για το πώς έχουν τα πράγματα. Να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Βερνιό, την Αντιπρόεδρο, η οποία μάλλον έχει καλά πράγματα να μας πει για τις επαγγελματικές ε, ε, δεξιότητες και την αμοιβαία αναγνώρισή τους. Μάλλον είναι καλά τα νέα. Ναι, μπορώ να σας πω ότι έχουμε καλά μαντάτα μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο αυτόν που θεωρούσαμε ότι θα είναι τελευταίο και πράγματι ήταν ο τελευταίο την περασμένη Τετάρτη. Νομίζω το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί στο Κοινοβούλιο και ευχαριστώ όλου που είστε παρόντε και το Κοινοβούλιο λέγω πραγματικά δώσαμε ευρωπαϊκό όραμα στις επόμενες γενιές. Όλοι κατέβαλαν καλές προσπάθειες και είμαι ευτυχέστατη γι' αυτό. Να σας πω εν συντομία ποια είναι τα κρεμή σημεία Όσον αφορά το επαγγελματικό τομέα, έχουμε ε, καλές προθεσμίες όσον αφορά και περιορισμό, περιορισμή παράταση των προθεσμιών να χρειάζονται συμπληρωματικέ πληροφορίε και αυτό δικαιολογείται και εγγυηθήκαμε να λάβουμε υπόψη τι απόψει των διαφόρων επαγγελματικών τομέων πριν ετοιμάσουμε αυτή τη χάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι το εργαλείο αυτό είναι ένα εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και είναι πολύ σημαντικό για του νέου που καλούνται να πάνε να δουλέψουν αλλού. Όσον αφορά τη μερική πρόσβαση, ένα κράτο μπορεί να αρνηθεί αυτή τη μερική ε, πρόσβαση και για λόγου εθνική ασφάλεια, αλλά όσου έχουν αυτόματη αναγνώριση, αυτό του αφορά. Όσον αφορά το καθεστώ το γενικό, όσον αφορά του παρόχου υπηρεσιών, δεν υπάρχει παρέκκληση αλλά χρειάζεται να υπάρχει πρώτερη επαγγελματική ερμηνεία και για τις διαφορετικά, διαφορετικά επίπεδα κατάρτισα κάτι μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν κάποιον που έχει χαλότερο από το bachelor αν απαιτείται ένα master. Αλλά τα κάτι μέλη έχουν περισσότερες δυνατότητες να έχουν ευελιξία για να επιβάλλουν μέτρα αντιστάθμισης. Και έχουμε εγγυηθεί ότι τα τεστ πρέπει να γίνονται εντός πολύ σύντομης προθεσμίας μετά την απόφαση της αρχής υποδοχής τουλάχιστον εντό εξαμήνου και όχι παραπάνω. Όσον αφορά τη συνεχή κατάρτιση, τα κάτι μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι όλοι οι επαγγελματίε θα πρέπει να τη χάνουν αυτόματη αναγνώριση που θα μπορούν να ενημερώνονται οι δεξιότητέ του μέχρι ότι τη συνεχού ε, επαγγελματική ανάπτυξη. Είναι σημαντικότατο αυτό για κάποια επαγγέλματα, κυρίω ε, για αυτά που δεν ακολουθούν συνεχή κατάρτιση. Για του γιατρού, η βασική πέδευση 5 ε, ετών και θα πρέπει να ε, δίνουν, να πετούν αν θέλουν μεγαλύτερη κατάρτιση πρέπει να μπουν διευκρινήσεις και χρειάζεται τεχνική ε, συνεδρίαση διευκρινιστή αύριο για τις διάφορες ιατρικές ειδικότητε. Μεθαύριο θα ζητηθεί για την ελάχιστη περίοδο ε, κατάρτισης, οπότε φαίνεται θα είναι τέσσερα χρόνια. Για τις νοσοκόμες δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το κείμενο, διότι η ΙΜΚΟ και το Συμβούλιο η Επιτροπή μας, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την ίδια θέση. Ε, σκληρή μάχη και τελικά καταλήξαμε σε κάτι καλό. Όσον αφορά τους κτηνιάτρους έγινε επικαιροποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Λοιπόν, πετύχαμε να περάσω 12 χρόνια η διδασκαλία και τις αρμοδιότητες και τις γνώσεις μέσω της αγωγής μιας αναφοράς στη φαρμακολογία για του φαρμακοποιού και να μπορούν να ασκούνται επάγγελμα ανεξάρτητα και έχουμε και ελάχιστη διάρκεια 4.600 ωρών περαιτέρω ε, πάνω από τα τρία χρόνια. Όσον αφορά του φαρμακοποιού δεν υπάρχει πρόβλημα. Η ενημέρωσή του ε, είναι κάτι που ζητήσαμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, το ίδιο για τους αρχιτέκτονες, με περισσότερες ειδικέ διατάξεις αφορά τι περιόδου μαθητείας, όπω ζητήσατε, στο κοινό πλαίσιο τη ε, κατάρτισης και εκεί είχαμε μεγάλες δυσκολίες και καταλήξαμε έχοντας να μείνουν οι κατεξοδότηση πράξεις λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες στις λεπτομέρειες. Αντίθετα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης αλλά από προκαθορισμένες συνθήκες καταφέραμε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο και να εφαρμόζεται επίσης τις ειδικότητε των διαφόρων επαγγελμάτων που αναγνωρίζονται αυτόματα. Το ζήτησαν οι επαγγελματίε αυτό. Όσον αφορά τις γλωσσικές δοκιμές, θα πρέπει να περιορίζονται στη γνώση μιας γλώσσας της χώρας υποδοχής και θα πρέπει να προσαρμόζονται τα τεστ ανάλογα με τον τόπο επαγγελματία θέλει να ασκήσει το επάγγελμά του και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μετά την αναγνώριση των ε, γνώσεών του. Όσον αφορά τη περίοδο μαθητείας, θα πρέπει να γνωρίζετε αυτόματα αν έχει γίνει σε άλλο κάτω μέλο η περίοδο μαθητείας και να λαμβάνετε υπόψη αν γίνεται σε τρίτη χώρα. Ε, οι στόχοι και το περιεχόμενο τη περίοδου μαθητείας θα πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων γραπτό. Όσον αφορά το μηχανισμό συναγερμού, λοιπόν, ε, υπάρχουν αναγκαία χέγγια Τέλος, όσον αφορά κατεξουδότηση πράξης για την αυτόματη αναγνώριση, επανεσύχθησαν αυτές οι πράξεις για την επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τις γνώσεις και τις εξιότητε, για τα αναγνωρισμένα επαγγέλματα που αναγνωρίζονται αυτόματα, εκτός από το νέο κατάλογο των γνώσεων για τις, ε, και τους νοσοκόμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι λιγότερο περιορισμένη για την θέτηση των πράξεων αυτών, γιατί η παρούσα οδηγία προέβλεπε ότι αυτές οι τροποποίησεις δεν θα έπρεπε να έχουν καμία συνέπεια όσον αφορά τις αρχές της νομοθετικής μιας χώρας, κάτι που μπορεί να εμποδίσει την πράξη κάθε προσαρμογή, ακόμα και μικρής εμβελίας. Ε, ενισχύθηκε και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, κυρίως όσον αφορά τις νέες διατάξεις και για τους νέους καταλόγους των διαφόρων γνώσεων των νοσοκόμων των νοσηλευτών και νοσηλευτιών. Ε, λοιπόν, καταλήξαμε σε καλά αποτελέσματα, σχεδόν αναπάντεχα, τουλάχιστον πολύ ικανοποιητικά σε σχέση με την εντολή που είχα την καλοσύνη να μου αναθέσετε. Ε, εκτός, δεν ξέρω αν υπάρχουν σκιώδεις εδώ, θα ευχαριστήσω τους σκιώδεις ηγητές για την θετικότητα θετικότατη συνεργασία που είχαμε. Χάρη στη δουλειά λοιπόν που κάναμε όλοι μαζί ε, και τα τι θεσμικά όργανα, πετύχαμε αποτελέσματα και η Ιρλανδική Προεδρία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τα ζητήματα και ήταν αποφασιστική η ενίσχυσή της. Ελπίζω ότι αυτή η ανάγνωση που θα κάνετε κατά την περίοδο ψηφοφορίας 9 και 10 Ιουλίου θα πάει καλά και βασίζομαι στην εμπιστοσύνη σας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον τρόπο που προεδρεύσατε των συζητήσεων στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ηγηθήκατε και τα αποτελέσματα πετύχατε πάρα πολύ καλά. Έχετε κάποιες ερωτήσεις για την Μπερναντέτ. Λοιπόν, τυπική διαδικασία είναι ότι περιμένουμε ο έγγραφο της Ενδικής Προεδρίας να επιβεβαιώσει ότι θα δεχτεί το κείμενο το Συμβούλιο. Ε, ελπίζω ότι αυτό θα το λάβουμε πριν τη συνεδρία επόμενης εβδομάδος και εν τη αυτή περιπτώσει θα τεθεί το θέμα υιοθέτηση του τελικού εγγράφου και θα μπει στην ημερήσια διάταξη προ έγκριση από την Επιτροπή και ανάλογα με τη θεσιμότητα τελικού κειμένου στι διάφορε γλώσσε για την Ολομέλεια. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου για επίσημη, διαδικασία, για επίσημη έγκριση. Ε, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η Επιτροπή ξεκίνησε τι εργασίε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση το 2009 δημιουργώντα μια ομάδα προβληματισμού ετοιμάσαμε δική μας έκθεση είχαμε επίσημε διαδικασίες που ετοιμαστήκαμε άριστα και φαίνεται ότι κάναμε δουλειά, φαίνεται στα σημαντικότατα αποτελέσματα την μεταρρύθμιση που θα γίνει να είναι πολύ καλύτερη η αμοιβαία αναγνώριση και θα είναι υποφελής για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ την Περνατέντη και τους άλλους. Προχωρώντας λοιπόν, εντάχει, δύο σημεία να αναφέρω. Να σας ενημερώσω ότι φτάσαμε σε συμφωνία όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής και τη σχετική οδηγία ε, χρειάστηκε χρόνος για να δούμε ποιες θα είναι οι, οι κατεξοδότηση πράξεις και διάφορες εφαρμοστικές διατάξεις. Υπήρξε συμφωνία, θα παρουσιαστεί το κείμενο αύριο για ψηφοφορία και λάβουμε και επιστολή από το Συμβούλιο που επιβεβαιώνει ότι δέχεται το κείμενο. Ευχαριστώ όλους λοιπόν για την υπομονή σας, διότι χρειάστηκε πάνω από ένα χρόνο για να φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Η κυρία Ρόιτεβα έχει ετοιμάσει μια έκθεση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο περίπλοκη, αρκετά περίπλοκη έκθεση, ως γνωρίζετε. Και ξέρω ότι ήθελε να είναι εδώ η ίδια, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Με... Μου ζήτησε να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Θα θυμόσαστε ίσως ότι ευθυγραμμίζονται εδώ ε, διάφορες οδηγίες με νέα προσέγγιση. Έπρεπε να επικαιροποιηθούν με τις διατάξεις συνθήκης της Αβώνας, αλλά χρησιμοποίησαν την ευκαιρία αυτή ούτως ώστε οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτών των μέτρων να ξεκαθαριστούν. Είχαμε οκτώ συγκεκριμένες οδηγίες που εξετάστηκαν, τεχνική φύσης τα θέματα, ε, τα δοχεία πίεσης, ε, ανελκυστήρες, ε, όργανα μέτρησης κλπ. Δεν εδώ σε λεπτομέρειες. Συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο επί όλων των σημείων και θα υπάρξει ευθυγράμμιση με το πακέτο 2008 για αγαθά. Πολλοί είχατε συμμετάσχει και στην πρώτερη θητεία της Επιτροπής και υπήρξαν και συγκεκριμένες απαιτήσει για τους ανελκυστήρες. Διότι είναι σημαντικά θέματα αυτά για την υγεία και την ασφάλεια και συμφωνήσαμε το πώς θα ακολουθηθούν οι εφαρμοστικές διαδικασίες, ποιος θα είναι ο ρόλος των επιτροπών, καθώς και πώς θα διαφυλάξουμε το δικαίωμα πρόσβασης εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρία εργασίας συνεδριάσεις που εξετάζουν όλα αυτά τα νομοθετικά στοιχεία. Γνωρίζετε πολύ ότι είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι σημαντικότατο να παρακολουθείτε η θέσπιση της νομοθεσίας και το πώς εφαρμόζονται τα νομοθετικά μέτρα. Η ε, κυρία Ρόιτεβα με τα χαράς σας, υποστη... σας παρουσιάσετε την πρόταση, προτείνει να τη στηρίξετε και θα πρέπει σύντομα να καταφτάσει και επιστολή της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας να επιβεβαιώνει όλα αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις, όχι, και αυτό για ενημέρωση για τα πρακτικά πάμε σε δύο άλλες οδηγίες όπου εξάγονται ακόμα διαπραγματεύσεις και προβλέπονται δύο συνεδριάσεις πριν το τέλος του μηνός οπότε θα ξεκινήσω με τον Μάρκ Ταραμπέλα να μας ενημερώσει τι γίνεται για το θέμα των δημοσίων προμηθειών και μετά το επόμενο θα είναι τι διάφορε άδειες και χωρίσεις. Ο Μάρκ Ταραμπέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, μόλις δύο νέες συνεδριάσεις ε, προβλέπονται 25 Ιουνίου 2 ε, με 5 για τις ε, δημόσιες προμήθειες και με και, και 10 με 11 το βράδυ και επίσης υπάρχει άλλη μία συνεδρίαση 21 Ιουνίου κοινή και για ε, τις δημόσιες αγορές και για τις παραχωρήσεις. Ε, στις 13 Ιουνίου είχαμε μία ακόμη τέτοια συνεδρίαση μεταξύ του Φιλίπ Ζουβάν και εμού και βέβαια ήταν και σκιώδης εισηγητές παρόντος σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και τις παραχωρήσεις. Ε, τέσσερα βασικά σημεία συζητηθήκαμε. Συζητήθηκαν συνεργασία δημοσίου-δημοσίου, το άρθρο 15.2 όσον αφορά τις γενικές αρχές. Για την συνεργασία δημοσίου με δημόσιο μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο μετακινήθηκε πάρα πολύ στη θέση του με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό που σημαίνει είτε αναφορά στον κύκλο εργασιών είτε στον αριθμό των δραστηριοτήτων, στις δραστηριότητες για τον υπολογισμό του 80% μπορεί δηλαδή να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο ως συμβεβασμός ή ο κύκλος εργασιών ή οι διαδραστηριότητες, γιατί ο κύκλος εργασιών δεν είναι δυνατόν πάντοτε ε, να υπολογιστεί επακριβώς, οπότε αφήσαμε κάπως ε, ένα ποσοστό ευελιξίας. Ε, αυτό δείχνει όχι μόνο τη σημασία του συντονισμού δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά πρέπει να υπάρχουν και μονάδες μέτρησης για να υπολογίσουμε αποτελεσματικά το 80%. Στην παράγραφο 1α γνωρίζετε, εκείνη πρωτοπρότεινα στο Συμβούλιο, Το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ε, νομίζω ότι μάλλον είχαμε καταλήξει συμφωνία. Στην παράγραφο 4 και 4α για την οριζόντια συνεργασία είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι γιατί είδαμε ότι ε, διαγράφηκε το genuine ε, που αναφερόταν στη συνεργασία, όπως επίσης και την, το carrying out jointly their public services, service tasks and involving mutual rights and obligations of the parties. Αυτό διαγράφηκε τελικά και αυτό συνάδει βέβαια με την ομολογία και με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η έκφραση, αυτή η διατύπωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ε, προβλήματα για την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών. Όσον αφορά τώρα την υπεργολαβία, το δεύτερο θέμα μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι για ε, την ε, εξέλιξη της θέσης ε, του Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι το 41 στις παραχωρήσεις αλλά το 71 στις δημόσιες αγορές. Είχαμε ζητήσει κάτι τέτοιο εμείς με την δική μας ψηφοφορία στις 24 Δεκεμβρίου στις 24 Ιανουαρίου και 18 Δεκεμβρίου. Ε, προφανώς 24 Δεκεμβρίου δεν ψηφίζουμε γιατί έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, ε, στη 15.2, στο άρθρο 15.2... Υπάρχουν ακόμη κάποια επίμαχα σημεία, διαφιλονικούμενα, που δεν μας ικανοποιούν καθόλου. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 5, Μα φαίνονται λίγο περίπλοκα, μα φαίνεται λίγο περί, περίπλοκη η διατύπωση. Είναι λίγο πιο περίπλοκα αυτά που μας λέει το Συμβούλιο σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε εμεί συμφωνήσει στο, Κοινοβούλιο. Αν το Συμβούλιο θέλει ανακούφιση των υποχρεώσεων ε, του οικονομικού φορέα, από την άλλη επανισάγει κάποιους νέους όρους, ε, άρα βγάζει κάτι από τη μία και το προσθέτει στην άλλη. Το συμβιβαστικό κείμενο λοιπόν ε, ζητά τις πληροφορίες ε, όχι μόνο προς τον υπεργολάβο, ενώ το κείμενο του Κοινοβουλίου ζητά αυτή η πληροφορία να γίνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της υπεργολαβίας. Είναι λίγο ιδιαίτερη λοιπόν η κατάσταση που δημιουργείται και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να εφαρμόσουμε τους κανόνες που προσπαθεί να περιγράψει το Συμβούλιο. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε κάτι σαφές, ε, πολύ συγκεκριμένο, το οποίο να μην θεωρείται μόνο απλώς γραφειοκρατικό, αλλά να είναι αποτελεσματικό για την αύξηση της ε, ε, διαφάνειας σε ολόκληρη την αλυσίδα της υπεργολαβίας και ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει. Για την παράγραφο 6 τώρα του κεφαλαίου και αυτό το άλλαξε το Συμβούλιο, αλλά φοβάμαι ότι δεν έγινε προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά, γιατί η διατύπωση του Συμβουλίου λέει ότι τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη ε, μία υπεύθυνη αλυσίδα υπεργολαφίας πρέπει να εξασφαλίζουν το σεβασμό του άρθρου 15.2 εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερο ότι αναφέρεται το άρθρο 15.2 που λέει ότι η σημασία που, που δείχνει τη σημασία που δίνουμε στο 15.2. Αυτό μας ικανοποιεί, αλλά δεν ε, μπορούμε να είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί με αυτή την παράγραφο, έτσι όπως είναι διατυπωμένη και όπως την ερμηνεύει το Συμβούλιο, μπορεί να αυξηθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που έχουν ήδη κάποιους κανόνες αποφασισμένους και τους ζητούμε να, τις, να τους κάνουν αυστηρότερους ακόμα, ενώ τα σύστημα που δεν έχουν τέτοιου είδους σύστημα ευθύνης ε, μπορούν να συνεχίσουν να μην το έχουν. Οπότε είναι δύο, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι λίγο παράδοξο και μου φαίνεται και λίγο απαράδεκτο να σας πω την αλήθεια, εφόσον θέλουμε να έχουμε πιο αποδοτική και καλύτερη ενιαία αγορά. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο καλούς κανόνες που να ισχύουν για όλους. Γι' αυτό θα ήθελα το Συμβούλιο να λάβει υπόψη να ε, να επανέλθετε στην προηγούμενη διατύπωση της ε, παραγράφου 6 από το ίδιο το Συμβούλιο ή στη δική μας θέση ένα ελάχιστο τέλος πάντων ε, ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα, τις πιο κλειστές αγορές θέλει να καλύψει μια κατάσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν λέω ότι γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να το δεχθούμε. Είναι ότι απλώς ε, ε, αφορά μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ε, περίπτωση της κοινωνικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου και γι' αυτό ακριβώς δεν θεωρώ ότι το άρθρο αυτό λαμβάνει υπόψη επαρκώς μια γενικότερη θεώρηση που ε, πρέπει να έχουμε για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες. Γι' αυτό εγώ δεν ε, βρίσκω ότι είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Η πρόταση της Επιτροπής την οποία μελετήσαμε υπάρχει, προβλέπει κλειστές ε, αγορές και είναι το άρθρο 76α το άρθρο αυτό 76α που είναι καινούριο άρθρο πηγαίνει προς, προς μια σωστή κατεύθυνση ενώ το 76β ουσιαστικά παραμένει στην διατύπωση του 76α όσο έχει αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως αυτή την υποχώρηση μπορούμε να την κάνουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο για το Συμβούλιο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση από ό,τι φαίνεται ως προς αυτό. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ένα βήμα προς τη δική τους θέση, αλλά βέβαια το 76β πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ε, μην ε, επιτρέψουμε κάποιοι, κάποιες αγορές να μπλοκάρουν κάποιες άλλες και να μην επιτρέπεται σε κάποιους οικονομικούς φορείς μέσω αυτής της διάταξης να μπλοκάρουν τις δραστηριότητες άλλων. Αυτά ήθελα να σας πω χωρίς να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ούτως ή άλλως ε, τα έχουμε ξαναπεί. Ε, πρέπει να γίνει μία αναδιατύπωση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της εφαρμογής των συλλογικών ε, συμβάσεων, ε, κάτι το οποίο μας απασχολεί εμάς πολύ στην Επιτροπή μας. Θέλαμε να υπάρχει μία αναφορά σε αυτό το θέμα και να μην υπάρχει επιλογή. Ούτως ή άλλως, σε πάση περιπτώσει, το δουλέψαμε πάρα πολύ οι τρεις συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου ελπίζουμε να μας ε, επιτρέψουν ε, στο πλαίσιο ακόμα της Ιρλανδικής Προεδρίας να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να γίνουν και κάποιες προσπάθειες ακόμη και κυρίως από την πλευρά του Συμβουλίου προς τη θέση του ε, Κοινοβουλίου, γιατί και εμείς το κάναμε για να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα σε όλου του οικονομικού φορεί, ιδιωτικού και δημοσίου, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, κύριε Πρόεδρε, ε, ήθελα να προσπαθήσω να σα μεταφέρω με πολύ πιστότητα αυτά που έγιναν. Νομίζω ότι βοηθούν αυτά. Αλλά σαν πρόεδρος θεωρώ ότι πράγματι επιτυχάνεται πρόοδος, διότι καταφθάνουν κείμενα από το Συμβούλιο και συζητούμε δύσκολα πολιτικά θέματα. Φιλίπ Ζουβέν, έχεις κάτι να προσθέσεις και εσύ σου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω αυτό που λέει ο Πολ Βαλερή, ο ποιητής ο Γάλλος. Αυτό που είναι αληθές είναι ψευδές, αυτό είναι που είναι περίπλοκο, είναι κάτι που εμπαξιμοποιηθεί. Άρα δεν θέλουμε να μην είμαστε πολύ ε, απλοί από τη μία πλευρά και να μην έχουμε και ένα άχρηστο κείμενο λόγω περιπλοκότητας. Άρα θέλουμε ισορροπημένο κείμενο. Σε πρώτερε συνεδριάσεις ε, πάντα ήμουν πολύ αυστηρό έναντι του Συμβουλίου που είχε μια στάση ε, άκαμπτη. Διαπραγματευόταν όχι από την αρχική θέση αλλά από την ε, πρώτη πρόοδο που είχε κάνει το Κοινοβούλιο. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήμουν αυστηρό εχθέ με το Συμβούλιο και είμαι πιο χαλαρό σήμερα. Και θα πω ότι το Συμβούλιο άλλαξε πραγματικά τη στάση του και η Προεδρία κατέβαλε σημαντικέ προσπάθειε για να λάβει υπόψη τι θέσει του Ευρωκοινοβουλίου επί σημαντικότητα των θεμάτων. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν με αργού ρυθμού και άλλοι δύο τριμερεί διάλογοι έχουν συμπληρωματικοί 21 Ιουνίου και 25 Ιουνίου και ένας από αυτούς είναι, θα λάβει χώρα με κοινή συζήτηση με τους για τις δημόσιες προμήθειες. Να διατρέξουμε τα άρθρα τώρα. Τα εκκρεμή θέματα. Οι ορισμοί του, η του κατοφλίου. υπάρχουν διαφορές εκεί. Για το άρθρο 36 για τις εξαιρέσεις μπορούμε να βρούμε σε τεχνικό επίπεδο λύσεις διαδικαστικά έχει έγκαια και τα κριτήρια διανομής. Ξεκινάμε από πολύ αντίθετες θέσεις. Νομίζω ότι θα βρούμε όμως κοινή προσέγγιση για την τροποποίηση των συμβάσεων. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το κείμενο διερωτάται μάλλον το Κοινοβούλιο διότι το κείμενο θα επέτρεπε ίσως κάτι που δεν θέλουμε ε, να παρατείνονται εσαΐ οι παραχωρήσεις και δεν το θέλουμε αυτό και θέλουμε κάποιες ε, διευκρινήσεις. Θα τα καταφέρουμε πιστεύω. Ένα σημείο που δημιουργεί προβλήματα είναι οι τομικές εξαιρέσεις άρθρο 8 της οδηγίας. Το Συμβούλιο δεν έχει μεγάλα περιθώρια λιγμών, διότι κάθε χώρα έχει θέση του όρου για τομεακές αποκλήσεις και εξαιρέσεις, άρα είναι πολύ ετερογενής οι θέσει του πάνελ και τα περιθώρια λιγμών είναι πάρα πολύ στενά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το Συμβούλιο, το αιτήμα του Συμβουλίου σε, στα, στη σφαίρα γενική Συμφωνίας για τα μεικτέ συμβάσεις, άρθρο 18 και 19, για μεικτέ δραστηριότητε, μπορούμε εκεί κάπου να καταλήξουμε, για το άρθρο 11, για τις επιχειρήσεις που διασυνδέονται, μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία, άρθρο 11α, το είχαμε προτείνει στο Κοινοβούλιο εμεί αυτό το άθρο που διθετεί το συγκεκριμένο θέμα του ύδατο που είναι σημαντικό. Λοιπόν, θα πρέπει να όλοι να δώσουν τις απόψεις του και μπορεί να αλλάξει ανάλογα το κείμενο. Έχουμε ερωτηματικά και θέτω το ερώτημα για τον επόμενο τριμερή διάλογο. Να δούμε νομικά. Μήπως δημιουργούμε κάποιο νομικό τέρας. Μήπως κλείνει και ιδιωτικοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες. Η προσέγγιση. Θέλουμε νομική άποψη για το 11α. Για το 15 συνεργασία δημοσίου-δημοσίου. Ο Μάρκο το ανέφερε εκτενώς. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Καλά πήγαν τα πράγματα. Δυσκολίε για την οριζόντια συνεργασία είχαμε, κάποιες μικροδυσκολίε. Θα πρέπει ίσω να συζητήσουμε. για να πλησιάσουμε περισσότερο διατύπωση της, ε, την ομολογία του δικαστηρίου. Και έτσι το άθρο να έχει τα σωστά πλαίσια. Κοινωνικέ στοιχείες. Έχει σημειωθεί πρόοδο από πλευρά Συμβουλίου στην αρχή, δεν ήθελε τίποτα, αλλά τώρα δέχεται κάτι. Από μακριά έρχεται σε αυτή τη θέση. Πολύ πολύ μακριά. Και τώρα μας προσεγγίζει. Αξιοσημείωτο, πολύ αξιοσημείωτο. Η υπεργολαβία επίσης το κείμενο διαγράφει το μεγάλο τμήμα του όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε και στι παραχωρήσει από το Συμβούλιο. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Είμαι λίγο πιο αισιόδοξο από τον Μάρκ εκεί. Υπάρχει ακαθόδε θέμα που ο Μάρκ Ταραμπέλα το ανέφερε. Αυτέ τα κλειστά, του κλειστού τομεί, κοινωνικέ υπηρεσίε, οι προσεγγίσεις μας ίσως διαφέρουν. Ανησυχώ λόγω της διατυπώσεων άρθρου που δημιουργεί ιδιαίτερο καθεστώς για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πουθενά όμως δεν έχουμε καθορίσει αυτές τις κοινωνικές εταιρείες. Όταν στο κείμενο του Συμβουλίου λέει κοινωνική επιχείρηση είναι με επιχείρηση που έχει στόχο κοινωνικό ή για γενικό σε πνεύμα κοινωνικό κινείται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μεθεί το societal το γαλλικό στα αγγλικά Για το κόστος το 76β είναι λιγότερο επικίνδυνο από το 76α ε, που μπορεί να παρερμηνευθεί. Ήταν θετικότατη η θέση του Συμβουλίου αυτή τη φορά. Πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος ήταν κάπως αργός και δεν ολοκληρώσαμε όπως θα θέλαμε. Μας μένουν τα τέσσερα σημεία, τα σκληρά θα έλεγα, τα όρια, τα κατόφλια τα θέματα για τις παραχωρήσεις για δημόσιες προμήθειες, το παράρτημα 10 για τις κοινωνικές και ειδικέ υπηρεσίες. Η περίπτωση του ύδατος θα πρέπει να το καθορίσουμε και πέμπτο σημείο σας, για τις συμβάσεις για διάφορους κλειστούς τομείς, αλλά μπορούμε πιστεύω εν γέννη να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Καλώς, ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, τις παρουσιάσεις. Ελπίζω να είναι πολύτιμες αυτές οι παρουσιάσεις. Έχετε τίποτα σχόλια. Η κυρία Στάλλερ έχει το λόγο. Για διευκρίνηση. Επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει 21 και 25 Ιουνίου και για τα δύο θέματα, σωστά άκουσα, για τους δύο επόμενους τριμερείς διαλόγους. Ο πρόεδρος κατ' εξαίρεση γίνεται μια συνεδρίαση Παρασκευή πρωί που δεν συνηθίζεται διότι χρειαζόμασταν και άλλο χρόνο. Διότι όπως είπαν και οι συγητές, καταφθάνουν πολλά περισσότερα κείμενα το Συμβούλιο, με πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν. Είπαν και οι δύο ότι αρχίζουμε να μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες ενός περιπλοκότατου ζητήματος, αλλά θέλουμε να δούμε και τελικά ποιος είναι ο σκοπός των μεταρρυθμίσεων και το κείμενο θέλουμε να είναι εύληπτο και προσβάσιμο και για τις συμβαλόμενες αρχές και για τους εκείνους που αφορούν οι συμβάσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και να πω, μιλώντας εκ μέρους των δύο συγγητών και των σκιωδών, ότι αναθέσαμε μία μελέτη από τη μονάδα εξολογή συνεπειών για τι συνέπειε που θα έχει αυτή η πρόταση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τι συνέπειε θα έχουν και αλλαγέ. Και έχει δημοσιοποιηθεί το πόρισμα τη μελέτη, έχει αποσταλεί στο Συμβούλιο, μα βοήθησε νομίζω αυτό στι διαπραγματεύσει και αν κάποιο θέλει να διαβάσει το κείμενο μπορεί να ρίξει μια ματιά. Το λέω δημοσία διότι δείχνει ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις ε, να γίνεται επικαταμερισμός σε μικρότερα κομμάτια συμβάσεων και θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τις προμήθειες μέσω του διαδικτύου ε, διάφορα θέματα που προωθούμε Καλώς, ευχαριστώ όλους σας Άφησα να χρονοτριβήσουμε λίγο, ήταν πολύ σημαντικό να γίνει δημόσια αυτή η συζήτηση του θέματος. Θα προσπαθήσω τώρα να καλύψω κάποιοι από τη χρονική στέρηση. Πάμε στο επόμενο σημείο σχέδιο πρότασης ψηφίσματο που έχει υποβάλει η Επιτροπή για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το πλαίσιο ποιο είναι, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή επί δυόμιση χρόνια εργαζόταν με συναφή θέματα που αφορούσαν την ψηφιακή αγορά. Έγιναν διάφορες συνεδριάσεις ομάδων εργασίας κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και αρκετοί από εσά ε, συμμετείχατε ε, τακτικά όπως ο κ. Δεκάμπος υπό την ηγεσία του Παύλου Αρίας και διαφόρων άλλων μελών που συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ετοιμάσαμε ένα ψήφισμα, το Κοινοβούλιο ετοίμασε ένα ψήφισμα που θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου και καλέσαμε και διάφορες άλλες επιτροπές ε, που ενδιαφέρονται να μας δώσουν κάποιες ιδέες Είχαμε ύψη τη ποιότητα τροπολογίε που υπευλήθησαν την Επιτροπή Πολιτισμού και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Μεταφορών, καθώ και την Επιτροπή Απασχόληση. Και νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται έτσι. Η Επιτροπή Βιομηχανία και η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου επίση. Η Επιτροπή Βιομηχανία ετοιμάζει παράλληλα ένα ψήφισμα για θέματα που άπτονται τη ενιαία αγορά για τι τηλεπικοινωνίε. Όλα αυτά θα ομαδοποιηθούν και από ό,τι έμαθα και από τη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων τη περασμένη εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη το πρωί της Ολομελία του Ιουλίου να διεξαχθεί συζήτηση για την ψηφιακή ενιαγορά θα επικεντρώνεται επί των ψηφισμάτων μα. Είναι καλό λοιπόν που είμαστε σε τέτοια θέση για αυτό το ζήτημα, σε κυρίαρχη θέση. Θα πρέπει αύριο τυπικά να ψηφίσουμε το περιεχόμενο του ψηφίσματος υποβάλαμε ο Πάμπλο Αρίας μάλλον και εγώ με τη βοήθεια της It Χαρτ που τη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανε και με τον Γιάν Χάρα, όχι, με, με την κυρία Χάρα που έχει γονική άδεια και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο αν μας λείπει από το σπίτι υποβάλαμε ψήφισμα και τροπολογίες έχουν υποβληθεί Πρέπει να εξετάσουμε τις τροπολογίες άλλων επιτροπών και να τις ψηφίσουμε αύριο. Ετοιμάσαμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν διανεμηθεί για να ενοποιήσουμε διάφορα τμήματα, διάφορα στοιχεία δικών μας τροπολογιών και επιτροπών άλλων που υπέβαλαν τροπολογίες και ελπίζω ότι θα εγκρίνετε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες και έχει ετοιμαστεί κατάλογο ψηφοφοριών που θα αναφέρεται σε όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση εκ μέρους του Παύλου Αρίας που δυστυχώς δεν παρίσταται ε, είχε υποχρεώσεις λοιπόν κάνω μια παρουσίαση εκ μέρους του σας ε, συστήνουμε να ψηφίσετε αυτό το πακέτο θέλω να ακούσω τυχόν σχόλια πριν πάμε αύριο για την ψηφοφορία ξέρω ότι ο Αντένιο Ντεκάμπος θέλει να σχολιάσει και είναι και σκιώδης και θα του δώσω το λόγο και σε οποιονδήποτε άλλον επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση είναι πρόσδεκτος. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Αντώνιο Κορία Κάμπους. Σας ευχαριστώ Μάκομ. Το κείμενο των συναδέλφων Παύλο Άρια και Μάκομ Χάρμπορ είναι πολύ περιεκτικό και πλήρες και αναφέρθηκε και στα κύρια συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας για την Ψηφιακή Αγορά, τον τρίτο κύκλο επαφών που συνήλθε πέντε φορές από την αρχή του έτους παρουσιάσαμε νέα τροπολογίες όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση κάποιων θεμάτων του κειμένου. Συμπεριέλαβα στα αρχικά σχόλια την αναφορά σε ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενιαία πράξη της επιχειρήσης και την ε, διαχείριση καθώς επίσης και για την ενιαία πράξη όσον αφορά την, τους υπολογισμούς cloud computing και τα προτερήματα όσον αφορά την ολιστική προσέγγιση, όσον αφορά την ανάπτυξη του, της ψηφιακής αγοράς. Επίσης την αμεροληψία και ουδετερότητα του διαδικτύου, το κόστος περιαγωγής, την αναζήτηση λύσεων όσον αφορά την e-procurement, ε, ηλεκτρονική προμήθεια, ηλεκτρονικές αγορές και με τη μορφή αυτών των τροπολογιών για το κείμενο ουσιαστικά έχουμε συνολικά ε, πολλές τροπολογίες ε, από διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες και 47 παρεμβάσεις από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες όσον αφορά την αποσαφήνιση θεμάτων στο κείμενο. Οι τροπολογίες από τις άλλες ε, κοινοβουλευτικές ομάδες και τις άλλες επιτροπές δεν δημιουργούν, δεν δημιουργούν προβλήματα και είμαστε σύμφωνοι με τους συμβιβασμούς, με τις συμβιβαστικές λύσεις. Έχουμε ένα πρόβλημα με την ε, τροπολογία 51 της Επιτροπής Γιούρη Νομικών Υποθέσεων που προσεγγίζει το θέμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Πώλησης και τοποθετείται για το ότι θεωρεί ότι η Σύμβαση Πώλησης είναι μια πρωτοβουλία λέει απόλυτα αναγκαία και θετική πρωτοβουλία πράγμα που ακόμα βρίσκεται υποσυζήτηση και υποανάλυση αυτή τη στιγμή. Η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα δεν δέχεται αυτή την αναφορά να γίνεται έτσι σε σχέση με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή πριν από την 8η Ιουλίου. Οπότε τότε θα συζητηθεί η κοινή πρόταση ΕΝΒΙ και ΙΝΚΟ σε σχέση με την πρόταση Γιούρι για την, ε, δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πολίσεων. Και για αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς είχαμε προτείνει ότι η καλύτερη λύση θα ήταν ή απλά να μην συμπεριληφθεί αυτή η τροπολογία και να μην ψηφιστεί που είναι το πιο, το πιο σταθερό επιχείρημα θα έλεγα, το πιο θεμητό επιχείρημα. Το περιεχόμενο στις 8 Ιουλίου από αυτού του θέματος θα συζητηθεί. Είναι να απόσχουν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες και να αποφύγουμε έτσι την μετατροπή αυτού του θέματος, δηλαδή ενός εξαιρετικού εγγράφου, σε ένα θέμα κατακαιρματισμού και διχασμού, πράγμα το οποίο δεν θα το θέλαμε. Ευχαριστώ. Okay, well, Καλώς. Ίσως αυτό μπορεί να προκύψει πριν ψηφοφορία αύριο. Λοιπόν, πώς τα βλέπω εγώ. Εν γέννη, όταν ένα θέμα είναι ευθύνη συγκεκριμένη επιτροπή, δεν προτείνουμε να ψηφίσουμε, το δεχόμαστε ανευ διότι ήδη ψηφίστηκε. Και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ψήφισε, είναι σαφέ. Προφανώ αυτή η Επιτροπή είναι εν μέρη υπεύθυνη. Μία λύση είναι να ψηφίσουμε αύριο. Και βλέποντα τι θα πούν τα μέλη. Ίσως θα ήταν χρήσιμο το μεταξύ να έρθουμε σε επαφή με τους εισηγητέ για τον κοινό ευρωπαϊκό κανόνα για τι πωλήσει, αν συστήνουν να απόσχουμε, τότε όλοι μπορούν να απόσχουν ή να καταψηφίσουν. Αυτός είναι ο δημοκρατικότερος τρόπος, αντί να αποφασίσουμε σήμερα. Να στείλουμε email σήμερα το απόγευμα στους δύο εισηγητές και να ζητήσουμε είτε αυτοί να πάρουν το λόγο ή κάποιος εκ μέρους τους αύριο πριν την ψηφοφορία και να μας πούν τι επιθυμούν να κάνουμε. Χαίρομαι που μας υποστηρίζετε εν γέννη. Άλλος Ο κ. Άγκστρομ θέλει να σχολιάσει. Κάποιο άλλο, Η κυρία Στάιλερ. κύριε, Βερχάιν. Η κυρία Γκάλερ. Ο κ. Άγκστρομ πρώτα απ' όλα. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Σχόλιο έχω. Συμβαστική, για τη συμβαστική τροπολογία. Δεύτερο τμήμα της πρώτης τροπολογίας πιστεύει ότι η δημιουργία τη ψηφική ενή αγορά μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν δίποτε διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών όσον αφορά την απασχόληση, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση τη ένδυα. Αν μπορούσαμε θα ήταν υπέροχο. Για να είμαι ειλικρινή, δεν περιμένω όλα αυτά να συμβούν μόνο από τη βελτίωση της ψηφιακής ενίας αγοράς, ίσως να υπερβάλλουμε λίγο εδώ. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω. Είστε απεσιόδοξο. Προσεκτική ήταν η διατύπωση. Ήταν το ψήφισμα τη επιτροπή απασχόληση. Μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν. Δεν λέει ότι θα ή θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν είναι σίγουρο, αλλά τα δημιουργεί τι συνθήκε Να, αν θέλετε ξεχωριστή ψηφοφορία, μπορείτε να το κάνετε αν δεν είναι αργά. Από εσά εξαρτάται. Η κυρία Στάιλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ εκείνου που ενδιαφέρθηκαν εκείνους που στην Επιτροπή δεν κατάφεραν να παραστούν στο εργαστήριο το ψηφιακό που κάναμε εδώ και μερικές εβδομάδες και τα διάφορα έγγραφα. Θα θέλαμε αυτοί οι συνάδελφοι να δουν τα έγγραφα. Ήταν χρησιμότατη η συζήτηση που έλαβε χώρα και ήταν η τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές. Και είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η δουλειά και ευχαριστώ και τους ηγητές και άλλους που συμμετείχαν. Εγώ ήθελα να πω ότι καλωσορίζω την αναφορά των ηλεκτρονικών βιβλίων στην παράγραφο 29 και 30 του πρωτοτύπου κειμένου και πόσο σημαντικό τομέα. Και θα πρέπει να αποφύγουμε, να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση όσον αφορά την πώληση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Αλλά το θέμα τη πρόσβαση των βιβλιοθηκών στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ένα θέμα. Και δεν θέλουμε η γνώση να έχει τιμή. Θέλουμε να μπορούν οι βιβλιοθήκες να προσφέρουν αυτά τα προϊόντα στους πελάτες τους. Και χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα περισσότερα να αναφέρονται στον πρώτο θέμα. Πράγματι πρόκειται περί υπηρεσίες, το αναγνωρίζω. Ίσως μπορούμε να βρούμε άλλο σημείο να αναφέρουμε αυτά τα ζητήματα όσο θα γίνονται πιο σημαντικά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το κόστος της να, λόγω του κόστου η γνώση να μην φτάνει στου πολίτε, γιατί θα έχουν πρόσβαση οι πολίτε στο μέλλον στα ηλεκτρονικά βιβλία. Πρέπει να δούμε προ το μέλλον. Καλό βήμα πρόοδο αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι την Πέμπτη στην Παρασ... στο Στρασβούργο θα το εξετάσουμε αυτό. Είναι τεραστία σημασία. Και ελπίζω περισσότεροι από την Επιτροπή μας να κάνουν την προσπάθεια να είναι παρόντες την Πέμπτη το πρωί και να συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Άλλος, άλλο σχόλιο. Ιούγκα Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ, εκ μέρους του συναδέλφου που δεν μπορεί να παρίσταται θέλω να πω λίγα λόγια Πρώτα απ' όλα, ο κ. Κίνκερκαρτ θέλει να πει ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και θέλουμε ε, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ψηφιακή αγορά. Γίνεται καλή δουλειά στην ομάδα εργασία. Είναι ευχαριστημένο που βλέπει οι τροπολογίε άλλων μελών τη ΣΥΜΚΟ ε, έχουν ληφθεί υπόψη. Δεν υπάρχουν συμβαστικέ για τι τροπολογίε ΣΥΜΚΟ, αλλά συμβαστικέ οι συμβαστικές είναι τεράστια, τεράστια πρόοδο σε σχέση με τις πρωτότυπες τροπολογίες. Καλώς. Όλοι είναι χαρούμενοι με τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Άλλος που έχει άλλα σχόλια. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευρία υποστήριξη. Όλα τα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν, μας υποστηρίζουν σε αυτό. Θα ψηφίσουμε αύριο και όταν θα έχουμε την ολομέλεια της Επιτροπής και τους ηγητές για τους ε, κοινέ ευρωπαϊκές πωλήσει θα δούμε τι θα κάνουμε. Η γραμματεία μου υπενθύμησε ότι απλή αποχή δεν αρκεί, διότι ουσιαστικά αυτό θα επέτρεπε να περάσουν οι τροπολογίε. Οπότε θα πρέπει να τις ε, καταψηφίσουμε αύριο, εάν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των συγητών, Από την άλλη μπορούμε να πάμε σε κατασυνήθιση ψηφοφορία, ό,τι θα αποφασίσουν οι ομάδες και να δούμε τι θα συμβεί. Ούτως ή άλλως θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, για τα πρακτικά να πω κάτι. Τετάρτη το πρωί θα είμαι στο Δουβλίνο, διότι η Ιρλανδική Προεδρία φιλοξενεί εκ μέρου τη Γενικής διεύθυνση για την Κοινωνία των Πληροφοριών, που εκπροσωπείται εδώ, όπω ο Νίκο Φόρτη, Λέω φιλοξενεί διήμερη διάσκεψη για την ψηφιακή ατζέντα και τη συνέλευση της ψηφιακή ατζέντα και την Τετάρτη πρωί θα συζητηθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά και μου ζήτησαν να προεδρεύσω στις συζητήσεις και προσβλέπω στην πρόθεση του ψηφίσματός μας σε αυτή την ε, συνεδρίαση και νομίζω ότι θα είναι και στο διαδίκτυο, θα γίνει web streaming. Αν θέλετε λοιπόν να ρίξετε μια ματιά Τετάρτη πρωί και να δείτε συζητήσει νέα ψηφιακή αγορά θα είναι στην ε, στο σελίδα της Γενικής Διευθύνσεως για την Κοινωνία των Πληροφοριών και μπορείτε να στείλετε Twitter μηνύματα θα μου διαβιβαστούν γιατί θα είμαι ο πρόεδρος της συνεδριάσεως. Όποιο παρακολουθεί λοιπόν στο διαδίκτυο και θέλει να συμμετάσχει στην Τετάρτη πρωί συζήτηση τη Γενική Διευθύνσεω για την Κοινωνία των Πληροφοριών και την ε, αρμόδια συνέλευση, είστε πρόσδεκτοι να συμμετάσχετε. Πάμε λοιπόν σε άλλη πρόταση που ενδιαφέρει πολύ τη συνέλευση για την ψηφιακή ατζέντα, για το ψηφιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής, ο κύριος Μάντερς, ο οποίος είναι απασχολημένος ε, διαπραγματευόμενος στο περιεχόμενο, όταν επιστρέψει στο κάθεσμά του θα μας το παρουσιάσει και αφορά το θέμα του την οδηγία για συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής διευθυνσής συγγενικών δικαιωμάτων και χορήγηση αδειών πολλαπλής ιδιωτικής εδαφικής ισχύω Έχουμε 242 τροπολογίες συνολικά. Είναι μια ευκαιρία να τις συζητήσουμε και να εξετάσουμε και τις συμβαστικές πριν την αυρινή ψηφοφορία. Θα δώσω το λόγο στον Τουάν Μάντρες, μάλλον να παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με χαρά έλαβα αυτές τις τροπολογίες. Νομίζω είχαμε μια επικοδομητική προσέγγιση για την εξέβρεση 44 συμβαστικών τροπολογιών κατά το μάλλον ή τον ελπίζω, πιστεύω ότι θα γίνουν δεκτές από όλους. Κάποιοι δεν μπορούν βέβαια να συμφωνήσουν όπως συμβαίνει πολλές φορές. Χαίρομαι για το ότι η συνάδελφος είναι παρούσα και ότι θα μπορούσε να δεχτεί κάποιες από αυτές τις τροπολογίες. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ιδιοκτητών πνευματικών δικαιωμάτων, να υπάρχει η δυνατότητα σαφής, σαφούς ε, εξόφλησης ε, υποβολής εμβασμάτων. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί και στους συμβιβασμούς και για τον ανταγωνισμό για την ενιαία εσωτερική αγορά που θα εμπλέκεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, διότι εργαστήκαμε σκληρά για αυτή τη γνωμοδότηση. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι είχαμε εμπλακεί και θέλαμε να βελτιωθεί η κατάσταση, όπως πρότεινε η Επιτροπή, να υπάρξουν βελτιώσεις. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες βέβαια που θα μπορούσα να τοποθετηθώ επ' αυτών. Ελπίζω όμως ότι η συμβιβαστική τροπολογία 17 που χρειάζεται κάποια περαιτέρω συζήτηση, όμως βρισκόμαστε στις 12 παρα 5 για την διατύπωση, για τα δικαιώματα τέλος πάντων πνευματικής ιδιοκτησίας και ελπίζω ότι θα υπάρξει υποστήριξη για την πρόταση και θα υπάρξει συμφωνία τελικά για να μπορέσουμε να εξεύρουμε τη σωστή διατύπωση. Είναι ένας συμβιβασμός προς αυτή την κατεύθυνση δηλαδή αυτός. Το ΕΛΚ τώρα. Και για την διαπραγμάτευση που έγινε. Δεν δέχονται την συμβαστική τροπολογία 41. Προτιμούν την αρχική τροπολογία του κυρίου Φαντεκάμπ. Η 43 αφορά υπολογισμούς. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε στο συμβιβασμό ότι θα υπάρξει μια εναλλακτική δυνατότητα προβλημάτων ή τριβών για την, να αποφασιστεί αν θα είναι δίκαια η έκβαση ή όχι. Ίσως όμως αύριο κατά τη διάρκεια της ε, ψηφοφορίας θα καταλήξουμε να δούμε αν έχουν πιστεί κάποιοι ή όχι, αν έχει πιστεί ο Μίγυρης. Και κατά το μάλλον ήταν για την υποστήριξη γενικά όλων των συμβαστικών τροπολογιών. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες δικαιωμάτων, αλλά και πάλι, ιδιαίτερα για τη συμβαστική τροπολογία 17, αν θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε την λέξη works, τότε θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα θετικό συμβιβασμό. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλου και τα μέλη της Επιτροπής ε, και όλοι είχαν εμπλακεί. Ελπίζω ότι αύριο θα τα καταφέρουμε. Η γνωμοδότησή μας δηλαδή να μπορέσει να πείσει και να ασκήσει επιρροή σε σχέση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Με ικανοποίηση βλέπω ότι ο εισηγητής από πλευρά τη Επιτροπής αυτής είναι παρόν για να παρακολουθήσει και να τίνει ευήκονους σε αυτές τις παρατηρήσεις. Και αν αναγκαίο, αν, είναι, αν ακόμα μπορούμε και να διαπραγματευτούμε με αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και μπορούμε να εξεύρουμε έναν αναγκαίο συμβιβασμό μεταξύ των κοινοβουλευτικών μας επιτροπών. Ίσως όμως δεν χρειαστεί αυτό. Ευχαριστώ όλους. Προσβλέπω στην ψηφοφορία αύριο. Well, thank you very much for your work. Ψηφοφορία αύριο. Ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε και ευχαριστούμε και την κυρία Γκάλερ για το έργο της ως εισηγήτριας και θα έχουμε τώρα ένα γύρο παρεμβάσεων από τους κοιόδης εισηγητές. Προτού το κάνω θέλω να καλωσορίζω μια ομάδα επισκεπτών που έχει προσκληθεί από την κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ, ιδιαίτερα ενεργό μέλος από πλευρά της ε, περιφέρειας Μάισνερ. Εσείς μάλιστα δεν ήταν τόσο κακή λοιπόν η προφορά μου. Καλώς ήρθατε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε να ε, σας δώσει θετικά στοιχεία συζήτηση και από πλευρά ε, του ΕΛΚΑ ε, είναι παρούσα η κυρία που θα παρέμβει. Ποιο θα παρέμβει εξ ονόματο ε, των Σοσιαλδημοκρατών. Η κυρία Μακλάκιν είναι παρούσα για την συνέχεια τη συζήτηση. Εσεί έχετε τον λόγο πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που έκανε εξαιρετική δουλειά από τις τόσες πολλές τροπολογίες να καταλήξουμε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς που στο τέλος τέλος σε κάποιες τοποθετήσεις που είναι διαφορετικές σε κατευθύνσεις και τοποθετήσεις μπορεί να ε, συγκλίνουν οι θέσεις σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις που θα έπρεπε να γίνουν εδώ, ωστόσο όμως σε τέσσερα σημεία θα θέλα δύο λόγια να πω. Αφενός για την τροπολογία 17 για την αφαίρεση κάποιων στοιχείων ε, όσον αφορά την, ε, στο πλαίσιο του συμβιβασμού όπως όμως προανέφερες και πάλι εδώ θα υπάρξει μια δυνατότητα συμβιβασμού. Δεν είναι δυνατόν εμείς να τοποθετηθούμε κατά όσον αφορά την δυνατότητα αδειών για τον μη εμπορικό τομέα. Όμως δεν θέλουμε να υπάρξει υπερβολικός κατακαιρματισμός στην αγορά που ζητούσαμε και με τις άλλες τροπολογίες και με τους άλλους συμβιβασμούς να αποφευθεί αυτό. Αν αφαιρεθεί ο όρος works λοιπόν θα μπορούσαμε να δεχθούμε αυτό το συμβιβασμό. Για την τροπολογία 41 τώρα πρέπει ειλικρινά να πω η διατύπωση σε σχέση με την τροπολογία όπως εξευρέθη από πλευράς Φαντενκάμπ βλέπω ότι είναι μια σαφέστερη διατύπωση από ό,τι του συμβιβασμού. Ίσως υπάρχει εδώ η δυνατότητα να καταφέρουμε να εξετάσουμε αυτή την τροπολογία και ενδεχόμενα αυτή την τροπολογία Φαντενκάμπ να την εντάξουμε καλύτερα ή αυτή να δεχτούμε μέσω της ψηφοφορίας. Στον συμβιβασμό 43 που τον προανέφερες μόλις, πρόκειται λιγότερο εδώ για το ότι δεν θέλουμε να ε, διευκολύνουμε σε δυσκολίες να μπορεί κανείς να προσφύγει σε αυτό το φορέα ε, διαμεσολάβησης αλλά θέλουμε τον τρόπο υπολογισμών των τιμολογίων να γνωρίζουμε πώς γίνεται. Είναι κάπως δύσκολο αυτό γιατί και σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις ε, να αποκαλύπτονται τέτοιου είδους υπολογισμοί το σημαντικό είναι οι όροι για, αυτή την τιμολόγηση και να δούμε πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί, να καλυφθεί όταν υπάρχουν κάποια εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχεία. Αλλά για έναν υπολογισμό λογαριασμών ή τιμολογίων, εδώ δεν κάνουμε λόγο για μη εμπορικές δραστηριότητες, αλλά για κυρίως εμπορικές δραστηριότητες, εμπορικού χαρακτήρα. Και για να δούμε αυτή τη διαφοροποίηση σε σχέση με επιχειρήσεις, για την αποκάλυψη στοιχείων τιμολόγησης πρέπει να προσέξουμε, να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν σε ένα νομοθετικό κείμενο κάτι τέτοιο να ενταχθεί ή όχι και να μην είμαστε υπερβολικά, υπερβολικά αυστηροί ή περιοριστικοί γιατί δεν πρόκειται μόνο για κάποιου τύπου δραστηριότητες ή μονοπόλια αλλά για ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο θέλουμε να ενταχθεί. Για τον συμβιβασμό 31 έχουμε και κάποιες δυσκολίες και με αυτόν. Εδώ περί τίνος πρόκειται. Όχι, μια στιγμή η 31 ήταν εντάξει, έβαινε καλός. Εντάξει, λάθος μου για τον υπολογισμό όταν θα πρέπει να έχουμε εμβάσματα ή collective costs. Δεν ξέρω ακριβώς το τι εννοείται. Αυτό ήθελα να αναφέρω και στη συνάντηση των συντονιστών, των σκιωδών εισηγητών. Οι συλλογικές αυτές εταιρείες διαχείρισης όταν ε, θα πρέπει να καλύπτεται αυτό το κόστος, αυτό όμως μπορεί να γίνεται μόνο αν και όταν έχουμε περιόδους υπολογισμού που είναι σαφείς ε, για τον, την έναρξη χρονικά των υπολογισμών αυτών μέχρι ότου να κλείσει μια περίοδος. Δεν θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την τροπολογία. Θα έλεγα να μην υποστηριχθεί από την ομάδα μας. Κατά τα άλλα είμαι ικανοποιημένη με αυτά τα οποία καταφέραμε. Από πλευράς αρχής δώσαμε αρκετά στοιχεία για μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία των δικαιούχων έναντι αυτών των εταιριών με μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστερα και σαφέστερα συστήματα για τους χρήστες του διαδικτύου και τους κατόχους αδειών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης αυτών των αδειών, αδειοδότησης και ικανοποιούμε με, τις, ε, με τους συμβιβασμούς που εξευρέθησαν. Ίσως σε αυτά τα τέσσερα σημεία μέχρι αύριο μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Ή διαφορετικά θα ψηφίσουμε ώστε να ρυθμιστεί με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βερχάιν. Ο κύριος Άγκστρομ. Ε, Ευχαριστώ. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες συμβιβαστικέ που μου δημιουργούν προβλήματα. Well, to, start with. Ξεκινάω. Τροπολογία 3, αιτιολογική σκέψη 3. Καταρχήν, τα κράτη-μέλη πρέπει τρέπεται να επιβάλλουν περιορισμούς όσον αφορά αυτούς που κινούνται στον τομέα. Νομίζω ότι είναι κατά της ε, ιδέας, της, το πνεύμα της οδηγίας. Ποιο ήταν το πνεύμα. Οι, αυτοί οι φορείς που ενεργοποιούνται σε ένα κράτος μέλος μπορούν να κινούνται διασυνοριακά. Τροπολογία 3 και άλλε ε, τροπολογίες απαγορεύουν κάτι τέτοιο αφήνουν τα κράτη-μέλη να εισάγουν οσδήποτε περιορισμού. Άρα αντιβαίνει το πνεύμα της οδηγίας. Και διαφωνώ, δυστυχώς. Αυτές που έχω υπογράψει εγώ, τις συμβαστικές τροπολογίες, σίγουρα δεν υποστηρίζω την τροπολογία 7 και την αντίστοιχη τροπολογία 32 στα άρθρα αν μια εταιρεία δεν μπορεί να βρει τα, τους δικαιούχους για να δώσει τα πνευματικά δικαιώματα, 7 και 32 λένε ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να κρατήσει τα χρήματα εάν δεν βρουν το δικαιούχο και να τα βάλουν σε ένα ταμείο που διχειρίζονται αυτοί για οποιοδήποτε σκοπό. Και αντί να τα δώσει στο δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι κίνητρο για να αυτές οι εταιρείε συλλογή δικαιωμάτων να κλέψουν. Είναι πολύ κακή ιδέα. Είμαι κατά και υποστηρίζω τις αρχικές μου τροπολογίες. Τροπολογία 12. Ορισμός αυτών των συλλογικών εταιριών. Ε, εδώ μπερδευόμαστε όλοι, δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Πολύ αοριστή διατύπωση, ανοιχτή. ή οργανια... οποιαδήποτε οργάνωση, οποιοδήποτε άλλο φορέα. Πρέπει να το σκεφτώ. Το λέω ότι προβληματίζομαι. Είναι πολύ ανοιχτή διατύπωση. Τροπολογία 14 που έχω υπογράψει, που έχει το όνομά μου. Τι ήθελα να κάνω εδώ. Για το άρθρο 3F 14. Για τον καθορισμό των εισοδημάτων από από τα πνευματικά δικαιώματα. δεν μπορεί να συνεχίσει η συλλογική εταιρεία αυτό που έκανε τώρα να μαζεύει πολλά χρήματα, να τα κρατάει επί μακρόν και να μαζεύει τόκους. Θέλαμε να το λύσουμε αυτό στον ορισμό. Στην υπόλοιπη οδηγία μιλάει για τα εισοδήματα από τα πνευματικά δικαιώματα. Τροπολογία 17, λυπούμε, δεν μπορώ να την υποστηρίξω ούτε αυτή. Θέλαμε να δώσαμε στους κατόχους των δικαιωμάτων να χρησιμοποιούν τις ελεύθερες, να δίνουν άδειες, ελεύθερες άδειες, εδώ λέει το αντίθετο. Οι δικαιούχοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις άδειες για δημιουργικούς σκοπούς. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους κατόχους των δικαιωμάτων, όχι τις συλλογικές εταιρείε. Έχουμε τις εταιρείε από τη μια πλευρά και τους δικαιούχους από την άλλη. Οι δημιουργοί πρέπει να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Να μπορούν να αποφασίσουν πώς να αδειοδοτούν, πώς να χρησιμοποιήσουν τις άδειε. Ίσως είναι λιγότερο επικερδές για τις συλλογικές εταιρείε, αλλά συλλογή των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά εγώ είμαι με το μέρος των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Τροπολογία 30. Δεν μπορώ να τη δεχτώ ούτε αυτή προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι οι σοικές εταιρείε μπορούν να κρατήσουν τα χρήματα μέχρι δύο χρόνια. Είχαμε αρκετέ τροπολογίε που, που έλεγαν ότι έπρεπε να καταβάλω τα χρήματα εντό τριμήνου. Ο συμβιβασμό λέει ξανά ότι αυτέ οι εταιρείε μπορούν να κρατήσουν τα χρήματα μέχρι δύο χρόνια. Κάναμε ένα πλήρη κύκλο και αφαιρέσαμε την ουσία από τις τροπολογίες ε, και από το συμβιβασμό. Δεν υποστηρίζω λοιπόν κάτι τέτοιο. Και τέλος, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος, αρκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Να σας υπενθυμίσω απλώς ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν και από πολιτικές ομάδες, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη όλη η Επιτροπή να τις υποστηρίξει. και αν ε, δεν περάσουν αυτές οι τροπολογίες, οι ουσιαστικές ε, τροπολογίες παρόλα αυτά ε, μπορούν να ψηφιστούν. Κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τουάν Μάντερς για την πολύ καλή δουλειά του στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε κάποιες καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ιδιαίτερα ευγνώμων είναι για την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από αυτό το ε, νομοθέτημα, γιατί είχαμε πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Η συζητήση είχε προτείνει να τις συμπεριλάβουμε, αλλά τώρα τελικά συμφωνήσαμε ότι θα τις τις μικρές συλλογικές εταιρείες θα τις προστατεύσουμε από το υπερβολικό βάρος, όπως ας πούμε τη λειτουργία επίβλεψης. Επίσης θέλουμε να μπορούν οι συλλογικές εταιρείες να συνεργάζονται για να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την αδειοδότηση, ε, όπως επίσης και για την ε, ε, για τα τιμολόγια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια κοινή τέτοια βάση δεδομένων να είναι διαθέσιμη online ε, για το για τον καταπιστευματοδόχο, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι ε, μπορούμε να το ε, λύσουμε όπως αναφέρεται στη διατύπωση. Ε, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει επαρκής ευελιξία για τα κράτη-μέλη ίσως θα έπρεπε να το τονίσουμε καλύτερα, με περισσότερο, με μια κάπως διαφορετική διατύπωση. Πάντως εγώ υποστηρίζω το να υπάρχει ε, ε, άδεια εδαφικής ισχύω ε, για τα μουσικά έργα γιατί πιστεύω ότι Κάτι τέτοιο ε, θα βοηθήσει την πραγματική ψηφιακή ε, ενιαία αγορά ε, να ολοκληρωθεί και, και τους χρήστες αλλά και τους οργανισμούς συλλογική διαχείρισης δικαιωμάτων θα τους ικανοποιήσουμε όλους. Και τους μεν και τους δε. Μήπως θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Μήπως από τους σοσιαλδημοκράτες θέλει κάποιος να συμβάλλει στη συζήτηση. Δεν ε, ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει. Όχι. Ωραία. Να δώσω τότε το λόγο στον κύριο Μάντερς να συνοψίσει. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η πρώτη μου πρόταση, κατά τη γνώμη μου, ήταν η καλύτερη ε, στα δικά μου μάτια. Αλλά αν, θέλετε να, αν θέλουμε να υπάρχει πλειοψηφία, πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, προφανώς. Νομίζω όταν λέει ο συνάδελφος ότι ε, ε, ότι ο συνάδελφος Έγκστρομ ε, λέει ότι δεν συμφωνεί με 6-7 από τις συμβιβαστικές τροπολογίες, ότι δεν συμφωνεί με αυτές και θέλει να ψηφίσουμε τις δικές του, εντάξει, μπορώ να το αποδεχθώ κάτι τέτοιο. Ως εισηγητής εγώ θα ήθελα να βρούμε ως το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία. Και αύριο θα το δούμε πώς θα πάει, αλλά ελπίζω πραγματικά έτσι να πάνε τα πράγματα. Η κυρία Γκάλο μήπως ε, θέλει να ε, πάρει το λόγο, γιατί είστε και εσείς η συγγήτρια. Απλώς και μόνο να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Μάντερς για τη δουλειά του. Ε, βεβαίως λάβαμε υπόψη τη δουλειά του. Έχουμε λιγότερο προχωρήσει εμείς σε σχέση με εσά. Έχω μία ακόμη συνεδρίαση με τους κοιόδους συζητητές στις 19 Ιουνίου ημέρα 5η. Ε, ημέρα Τετάρτη και ε, την Πέμπτη το πρωί πρέπει να τις ε, συμβιβάσω όλες. Είναι 450 οι τροπολογίες, οπότε πραγματικά έχω πάρα πολλή δουλειά. Το πρόβλημα είναι τα χρήματα, πόσο θα τα κρατάμε, τι θα τα κάνουμε. Τα ίδια ζητήματα τίθενται και στη δική μας Επιτροπή. Όλοι συμφωνούμε για την ε, καλύτερη ε, διαχείριση, για την καλύτερη διαφάνεια των ε, εταιριών συλλογική διαχείρισης. Νομίζω ότι και εσείς και εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Όπως επίσης και με την άδεια πολλαπλή εδαφική ισχύω, κάτι το οποίο θα δώσει το δικαίωμα στον Ευρωπαίο πολίτη να ε, καταναλώνει πολιτιστικά αγαθά ε, πέρα από τα ε, σύνορα της χώρας στην οποία διαμένει. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, 9.45 θα ψηφίσουμε αύριο, σας το υπενθυμίζω να φέρετε και την ε, ηλεκτρονική σας κάρτα ψηφοφορία. Συγγνώμη, θα σηκωθώ λίγο γιατί έχει μου διάσει το πόδι μου. Συγγνώμη. Ελπίζω λοιπόν ότι οι συμβιβαστικέ αυτές τροπολογίες θα τύχουν υποστήριξη και στη δική σας ε, επιτροπή, κυρία Γκάλο. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη. Να ελέγξω όμως ποιο είναι εδώ. Στο 7 πρέπει να πάμε κανονικά. Ο κύριος Διγιόγκ όμως δεν έχει έρθει, είναι ο εισηγητής μας για αυτό το θέμα. Οπότε δεν ξέρω αν είναι κανείς άλλος από την ΚΟΥ εδώ. Εγώ λέω να διακόψουμε λιγάκι μέχρι να εμφανιστεί ο κύριος De Jong. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά και τους ε, επισκέπτες μας θα ήθελα να ευχαριστήσω. Όταν έρθει ο κύριος De Jong, θα αρχίσουμε την πρώτη μας συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Λιανικό Εμπόριο. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, γιατί έχουμε εδώ τους ε, βασικούς πρωταγωνιστές ε, για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να αρχίσουμε δηλαδή τη συζήτηση για μία έκθεση πρωτοβουλίας Επιτροπής μας, ε, που είναι η ανταπόκρισή μας στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχέδιο δράσης για το λιανικό προεμπόριο, το οποίο δικό μας θα λέγεται σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων. Κύριε Ντεγιόν, καλώ ήρθατε. Είναι και η κυρία Χάντζλικ εδώ που εκπροσωπεί την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, έχουμε τη συνάδελφο από τους ε, σοσιαλιστές ε, και ο Τουάν από ό,τι βλέπω θα εκπροσωπήσει τον κύριο Λόκεγκαρντ. Ή τέλο πάντων δεν ξέρω αν έρθει κάποιο άλλο από του φιλελεύθερου και εγώ θα είμαι σκιώδη συζητητή για τη δική μου ομάδα. Η Μαρία Ρέιμπιντα είναι εδώ από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ, ε, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με ζητήματα business to business. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ, μαζί με τους συναδέλφους σας από τη Γενική Διεύθυνση ε, Μάρκτ. Ε, θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον συνάδελφο Ντεγιόντ να μας πει τι θέλει να κάνει με αυτή την έκθεση. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ θερμά Μάκομ και ζητώ συγγνώμη για το ότι καθυστέρησα κάποια λεπτά. Πολλές συνεδριάσεις ε, διεξάγονται εκ παραλλήλου αυτό το απόγευμα. Αλλά αληθεύει είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό για την ΙΜΚΟ. Και νομίζω ότι έχουμε και παράδοση αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων με την έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ για παράδειγμα. Συζήτησα με την Άννα Μαρία γιατί στόχος μου είναι να δώσουμε συνέχεια με τη γραμμή που είχε υιοθετήσει η έκθεση Κοράτσα Μπίλτ έκανε ήδη υπέβαλε ήδη αρκετές σημαντικές προτάσεις και πρέπει να τις συγκρίνουμε τώρα με το πρόγραμμα δράσης και να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε την συνάφεια και συνεκτικότητα στις τοποθετήσεις μας με την περαιτέρω παραγωγή προτάσεων από πλευράς μας. Να έχουμε δηλαδή μια συνεκτική και συνεπίγραμμη, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε ε, σε όλα τα σημεία, είναι σημαντικό οι συζητήσεις να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που δημιουργήθηκε το πρόγραμμα δράσης και ε, υιοθετήθηκε η προηγούμενη έκθεση, άλλαξαν πολλά πράγματα. Είχαμε και την, την, την ε, κρίση και το λιανικό εμπόριο επλήγει ιδιαίτερα σοβαρά στην Ευρώπη τα κέρδη, τα έσοδα μειώνονται και ιδιαίτερα στον τομέα εκτός τροφίμων αλλά και γενικά. Και αυτά όλα δεν επεξηγούνται απλά και μόνο λόγω της μετακίνησης προς το διαδίκτυο. Όλο και περισσότερο είναι δημοφιλές πλέον σήμερα το διαδίκτυο και αυτό έχει και τις επιπτώσεις του στο τζίρο των επιχειρηματιών. Έχουμε και ε, καταστήματα τα οποία δεν έχουν υπηρεσίες διαδικτύου και οι επιδόσεις τους ε, δεν είναι και τόσο καλές. Έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και το πρόγραμμα δράσης. Από πλευράς έκθεσης ε, θα θέλαμε να επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα δράσης ώστε να προσαρμοστεί και να λαμβάνει υπόψη τα όσα τεκταίνονται στην οικονομία μας σήμερα. Να επικεντρωθούμε σε μικρά ανεξάρτητα καταστήματα και επιχειρήσεις. Αναφερθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση με ε, τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθούν οι δραστηριότητες αυτών των μικρών καταστημάτων. Αυτό ήταν μια τοποθέτησή μας. Ε, κυρίως τα μικρά μαγαζιά, τα μικρά καταστήματα είναι εκείνα τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από αυτή την κρίση σήμερα. Έτσι λοιπόν ακούσαμε από πλευράς Επιτρόπου ότι ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα και θα ήθελε να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων, αλλά δεν θα πρέπει να αναμείνουμε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση άμεσα. Προτού ε, εξαλειφθεί αυτός ο τομέας δραστηριοτήτων με αυτά τα μικρά μαγαζιά ε, συνολικά. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτά τα καταστήματα και να συνεχίσουν με τις δράσεις τους. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να διασφαλίσουμε την ε, πολυμορφία από πλευράς αυτών των ε, δράσεων και τα δικαιώματα να μπορούν οι καταναλωτές ε, να καλύπτουν τις ανάγκες τους ακόμα και όταν ε, ζει κάποιος σε ένα χωριό να μπορεί για παράδειγμα να διασφαλίσει ως καταναλωτής τα δικαιώματά του. Είναι σημαντικό και αυτό το οποίο αναφέρεται στην έκθεση ότι αυτός ο τομέας δεν είναι όπως άλλοι οικονομικοί τομείς δραστηριοτήτων διότι έχει μια ιδιαίτερη πολιτισμική και κοινωνική αξία. Έρευνα έγινε πρόσφατα που καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι η συχνότητα κοινωνικών επαφών μεταξύ ατόμων στην κοινωνία μας μειώνεται η συχνότητα αυτών των ε, επαφών. Δεν έχουμε πια ε, γραφεία ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών για παράδειγμα, ταχυδρομεία παντού, επίσης βιβλιοθήκες και έτσι εκτός εργασίας τους είναι σημαντικό να διασφαλίζονται οι κοινωνικές αυτές επαφές. Οι επαφές είναι πολύ σημαντικές για τις διατομικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ανθρώπων. Όμως όλοι αγοράζουμε σήμερα στο διαδίκτυο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, αυτό θα έχει μια αρνητική κοινωνική επίπτωση. Βλέπουμε τις επιπτώσεις όλων αυτών ε, των εξελίξεων και στην απασχόληση επίσης και ε, στο λιανικό εμπόριο έχουμε και ε, απασχολούμενους, απασχολούμενους με χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων ή ικανοτήτων, ε, άλλους με υψηλότερο, διτή προσέγγιση πρέπει να υιοθετηθεί. Ή θα δεχθούμε ότι αυτά τα μαγαζιά έχουν πλέον ξεπεραστεί και ανήκουν στο παρελθόν και το μέλλον θα ανήκει στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το μόνο που χρειάζεται είναι μεγάλα καταστήματα, μεγάλα κέντρα όπου μεγάλα μαγαζιά και καταστήματα θα δραστηριοποιούνται όπως shopping malls, μεγάλα κέντρα καταστημάτων ή θα προσεγγίσουμε περισσότερο και θα επικεντρωθούμε στην ενδυνάμωση των μικρότερων καταστημάτων. Εγώ θα ήμουν υπέρ αυτής της δεύτερης επιλογής. Πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και προσαρμογές. Δήμοι, κοινότητε, ε, αναφέρονται αυτά σε σχέση με την έκθεση. Υπάρχει μια δυνατότητα να δίνονται προτεραιότητε στα μικρά καταστήματα σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων στο Ρότερνταμ από το οποίο προέρχομαι, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα καταστήματα πάβουν πλέον να υφίστανται. Έχουμε επενδύσει με σημαντικές δράσεις και από πλευράς του εμπορικού επιμελητηρίου και από πλευράς ε, του κοινού με χρηματοδότηση ώστε να αναζωογονήσουμε και καταφέραμε να αναζωογονήσουμε αυτά τα ε, καταστήματα το να μπορεί κανείς να πηγαίνει σε ένα τέτοιο κατάστημα ώστε να ε, έχει κάποιες δυνατότητες παράδειγμα και να ε, κρατηθεί το επίπεδο αυτή τη κοινωνική δραστηριότητα. Σημαντικό είναι να υπάρχουν επιχειρηματίε που θα μπορούν να δημιουργούν το κατάστημά τους με προϊόντα τα οποία ίσως οι ίδιοι παράγουν ή παρασκευάζουν και να εντάσσεται το κατάστημά τους σε ένα τέτοιο δημοτικό επίπεδο ώστε να είναι θελκτικό κιόλα για τους καταναλωτές και να μπορεί να τους προσελκύει. Είναι παραδείγματα θετικών πρωτοβουλειών. Σε μια γειτονιά για παράδειγμα που αντιμετώπιζε δυσκολίες και καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εμπορική οδό με τέτοιες δραστηριότητες που θέλει προσελκύει πολίτες και καταναλωτές και στο Ρότερνταμ το είδαμε ότι το μεγαλύτερο κέντρο καταστημάτων θα δημιουργηθεί ε, εκεί πάρα πολύ πιθανότατα θα πηγαίνουν λοιπόν σε αυτή τη γειτονία και θα έχουμε και την ίδια πίεση που θα ασκείται και σε άλλες περιοχές. Δεν είναι λοιπόν ε, μια πάρα πολύ ε, συνεκτική και συνεπής πολιτική αυτή η οποία ακολουθείται σήμερα. Θα πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς στην προσπάθεια να διατηρήσουμε και να διασφαλίζουμε την ύπαρξη αυτών των μικρών καταστημάτων. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό το, στο οποίο αναφέρθηκε και η προοπτική του ε, δικαστηρίου, του 10, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν είναι μόνο το θέμα των ε, ε, αδειών για τέτοια καταστήματα, αλλά πρέπει πρέπει να δούμε και τον μοναδικό χαρακτήρα που μπορούν να έχουν αυτά τα μικρότερα καταστήματα. Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει κανείς ε, στην υποστήριξη αυτών των καταστημάτων. Μπορεί να υπάρξει επιδότηση για παράδειγμα ενοικίων ή μισθωμάτων γιατί διαφορετικά θα είναι υπερβολικά υψηλά τα μισθώματα για τέτοιου είδους καταστήματα και το βλέπουμε πολύ συχνά σαν αποτέλεσμα όλων αυτών στα κέντρα των μεγάλων πόλεων το ίδιο είδος ε, καταστήματος επαναλαμβάνεται και συναντάται κατ' επανάληψη ε, χωρίς να διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και σε ποιο βαθμό μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνεργασία όσον αφορά καταστηματάρχες ώστε να αναπτυχθεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς αυτών των καταστημάτων. Είναι σημαντικό να υπάρξουν ενώσεις καταστηματαρχών που θα επομίζονται την ευθύνη για ένα, μια ευρύτερη περιοχή. Να δούμε όμως ε, σε ποιο βαθμό αυτό έχει επιπτώσεις και στον ίδιο τον ανταγωνισμό και τα θέματα ανταγωνισμού. Υπάρχει εδώ και το θέμα της πολιτικής ανταγωνισμού. Σε ποιο βαθμό δηλαδή τα μικρά καταστήματα θα μπορούσαν να υποστηρίζονται από μια τέτοια πρωτοβουλία που θα αναλαμβάνεται από τους κατοίκους τέτοιων γειτονιών και πώς θα μπορούσαν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να υποστηρίζονται από τις κυβερνήσεις από τους ε, υπευθύνους από πλευράς κυβερνήσεων. Τι θα μπορούσε να γίνεται στον τομέα δηλαδή του λιανικού εμπορίου για να τονωθεί αυτό. Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν φαίνεται να προσέχουν ε, όλοι αυτό το θέμα. Το θέμα της ε, φοροδιαφυγής, για παράδειγμα, έτυχε ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά την εταιρεία Starbucks, για Starbucks στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πολλά μικρά καφενεία φυσικά στην Ολλανδία. Είναι διαφορετικού είδους καταστήματα αυτά. Πολλά όμως από τα απλά κανονικά καφενεία ε, χρεοκοπούν επειδή αναλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες η εταιρεία Starbucks και φοροδιαφεύγει κιόλας και επιπλέον. Βλέποντας λοιπόν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ θετικό. Προβλέπει διασυνοριακές δραστηριότητες και έχει και αυτό την αξία του. Θα έλεγα, η έκθεσή μου οπωσδήποτε θα υποστηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα τις συμπληρώνει και με διάφορα ξεχωριστά σημεία. Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης αφορά αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού. Εδώ ε, εφιστά την προσοχή μας σε μια καλύτερα λειτουργούσα αλυσίδα τροφικών ε, προϊόντων, ε, τροφική αλυσίδα. Ε, διατροφική αλυσίδα. Είναι σημαντικό αυτό διότι υπάρχουν και αθέμητες πρακτικές που συναντώνται μονομερείς αλλαγές για παράδειγμα όσον αφορά τις ε, αλλαγές τιμών και την αλλίωση της ε, ε, συμπεφωνημένης πολιτικής ε, τιμολόγησης και τιμών. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα αθέμητων πρακτικών. Όσο περισσότερο εμβάθυνα και εξέτασα αυτό το θέμα, τόσο περισσότερο κατέληγα στο συμπέρασμα ότι εθελούσιες, εθελοντικές συμφωνίες θα ήταν μια καλύτερη δυνατότητα από ότι δεσμευτικές ή επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Όχι ότι είμαστε εναντίον ενός τέτοιου πλαισίου, αλλά ε, βλέπουμε ότι βρίσκονται σε διαφορετική θέση οι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το εμπορικό πλαίσιο, διότι ο ανταγωνισμός, για παράδειγμα, ε, οδηγεί στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι θέμητα. Δεν είναι αναγκαστικό να καταλήγει κανείς στην ε, διαμεσολάβηση ή στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων του προσφεύγοντα ένα τέτοιο φορέα. Διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις από πλευράς του προμηθευτή. Δεν είναι λοιπόν αναγκαία αναγκαίο να ε, δρομολογούνται υποχρεωτικά ε, μονομερώς αυτές οι ε, δυνατότητες. Μία εθελούσιου, εθελοντικού χαρακτήρα τέτοια συμφωνία θα ήταν ίσως μια καλύτερη δυνατότητα. Να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας ώστε σε μια άτυπη βάση να μπορούν οι πολίτες να έρχονται σε επαφή με αυτόν τον φορέα. Ίσως κλαδικές οργανώσεις και ενώσεις να μπορούν να προσφεύγουν σε ένα τέτοιο φορέα για την εξέβρεση λύσεων και εναλλακτικών δυνατοτήτων. Αυτό θα ήταν ίσως σε μια καλύτερη προσέγγιση από μια άκαμπτη κανονιστικού χαρακτήρα ε, προσέγγιση. Και να δούμε κατά πόσον σε σχέση με την έρευνα που έχει γίνει και καταδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα είναι η διανομή ε, προϊόντων από μεταποιητικές ε, βιομηχανίες και εταιρείε. Εδώ υπάρχει εμπλέκονται και οι μικροί, ε, μικρής κλίμακας γεωργοί, τα προϊόντα των οποίων περνάνε στην αλυσίδα, την διατροφική αλυσίδα και τα οποία εμπορεύονται και μεγάλες επιχειρήσεις ή υπεραγορές. Αυτό δεν αποβαίνει προς όφελος λοιπόν υποχρεωτικά των ε, ε, αγροτών αλλά υπέρ των υπεραγορών. Αν δει κανείς λοιπόν το τι γίνεται με την προμήθεια αυτών των ε, υπεραγορών με τέτοιου είδους προϊόντα από μικροπαραγωγούς, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εμπλοκή σε αυτή την εθελοντικού χαρακτήρα ε, προσέγγιση. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Πρέπει να μπορούν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν. Αν δεν συμμετέχουν τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει διασύνδεση όλων των κρίκων της αγοράς και δεν θα καλύπτονται επαρκώς. Θέλω να υπαρκεστώ σε αυτά τα σχόλια. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην ε, ε, υπαχθούν εδώ υπερβολικά σχετικά πολλές νομοθετικές προτάσεις, αλλά προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Για τις υπεραγωγές, για τις υπεραγορές, με συγχωρείτε, έχουμε και το θέμα πολλές φορές ε, υπερτιμολόγηση. Θα έπρεπε να υπάρχουν συμφωνίες ε, ώστε να εξετάζεται η δυνατότητα επιπλέον 5% ε, στην τιμή πώληση των προϊόντων των μικρογεωργών Ίσως αυτό θα πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει κάτι παραπάνω γι' αυτό. Να αποφύγουμε να δημιουργηθούν μόνο ολιγοπολιακές ε, καταστάσεις. Αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο, ακόμα και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, θα ήταν δύσκολο σε μια περίοδο κρίσης να υπερασπιστεί κανείς ένα τέτοιο μέτρο αύξησης ε, των τιμών με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι τιμές σήμερα, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πλαίσιο ανεξέλεγκτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη εισαγωγή. Καλύψατε πάρα πολλά θέματα και χαίρομαι γι' αυτό. Υπήρξε και πράσινη βίβλος ε, για τις ε, θεμητές ε, εμπορικές πρακτικές, κάτι το οποίο πρέπει επίσης να το δούμε σε σχέση με αυτά που αναφέρατε. Ας αρχίσουμε με τους κοιόδης εισηγητές, να αρχίσουμε με την κυρία Χάντσλι και εκ μέρου της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πράγματι, η κυρία Κοράτσα Βίλτ ε, ζητά συγγνώμη για την απουσία της. Ε, μου ζήτησε να σας ε, ενημερώσω και να σας μεταφέρω κάποια από τα σχόλιά σας. Τα Στηρίζει λοιπόν, ε, χαιρετίζει το γεγονός ε, ότι το θέμα του λιανικού εμπορίου είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες ε, και πυλώνας της ενιαίας αγοράς, κάτι το οποίο δείχνει πόσο δεσμευμένοι παραμένουμε ως Κοινοβούλιο για την ενθάρρυνση του περιφερειακού εμπορίου και κυρίως σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο ενθαρρύνει τον κύριο Ντε τον εισηγητή, να λάβει υπόψη ε, όλα όσα έχουμε επιτύχει ως τώρα. Σε μία από τις εκθέσεις της, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ε, ανέφερε και η έκθεση είχε τίτλο ε, «Προς ένα δικαιότερο λιανικό εμπόριο». Ε, και κυρίως αναφερόταν στα θέματα B2B, ε, business to business. Έλεγε λοιπόν η έκθεση τότε της κυρίας Κοράτσα Μπίλντ ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντικές και θεωρεί ότι αυτή η έκθεση που θα εκπονήσουμε τώρα θα ε, βελτιώσει περαιτέρω τον τομέα του λιανικού εμπορίου και θα δημιουργήσει επικοδομητικό διάλογο ε, τον οποίο ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Πριν από τρία χρόνια είχαμε την ίδια συζήτηση όταν το λιανικό εμπόριο άρχισε να υπάρχει ε, στις προτεραιότητές μας για πρώτη φορά. Βλέπουμε πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πάει καλά το λιανικό εμπόριο, αλλά ε, δυστυχώς ε, περνάει η κρίση. Τα διατροφικά σκάνδαλα αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μας και ε, δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη διαφάνειας και όχι μόνο στον τομέα των τροφίμων όχι μόνο χαμηλές τιμές θέλουν οι καταναλωτές, θέλουν και ποιότητα. Ε, θέλουν να μπορούν να συγκρίνουν ε, τα συστατικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος και την ποιότητά του. Η κυρία Κοράτσα Μπιλ θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο συζήτησης, ειδικότερα ως προς τις, ε, τα ιδιωτικά σήματα και τις καινοτομίες. Πώς θα αναπτυχθούν αυτά τα ιδιωτικά σήματα. Τα θέλουν οι καταναλωτές μας, ε, δίνουν πραγματικά πλήρη ή μεγαλύτερη εικόνα έστω στους καταναλωτές μας άποψη της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ είναι ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ακόμη ανησυχίες σε σχέση με ε, την πρόσβαση σε μικρά ε, καταστήματα λιανικής πώλησης, κυρίως ε, σε αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο των μεγάλων εμπορικών κέντρων και της επιλογής που δίνουν αυτά. Πρέπει να, να θυμόμαστε ότι ε, η ανάπτυξη των πόλεων ε, είναι πέρα από την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε θέματα διοδότησης ε, ή σχέδια τοπικής ανάπτυξης. Είναι όμως πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε παρκείς συνθήκες για ελεύθερο, δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό, όπως επίσης και ελευθερία επιλογής για όλους τους καταναλωτές. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ είναι της απόψεως ότι πρέπει να ευστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας ε, στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ειδικότερα στις περιπτώσεις B2B, να παρακολουθούμε τη διαδικασία της αυτορύθμισης. Τα τελευταία χρόνια κάναμε ένα μεγάλο άλμα προς έναν πιο επικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των ε, παραγόντων που τώρα είναι υπεύθυνοι για ε, μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ε, δικαιοσύνη στο λιανικό εμπόριο. Περιμένουμε να δούμε Πού θα ε, καταλήξουν όλα αυτά. Η ελευθερία της ε, κυκλοφορίας, όπως επίσης ε, και το επιχειρηματικό πνεύμα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Παρόλα αυτά, όλα, όλοι οι παράγοντες πρέπει να επιμείνουν σε υπεύθυνες και διαφανείς πρακτικές. Και ελπίζω η έκθεση αυτή να βοηθήσει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φάρει τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ακόμη στο, ε, στο λιανικό εμπόριο θα είναι ε, ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και το τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Μπορεί να είναι ένας τρόπος ε, να δεσμευθούν ε, όλα τα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό η κυρία Κοράτσα Μπίλτ περιμένει στενότερη συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, αναμένει εναγωνίως επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές και είναι σίγουροι ότι μπορεί να υπολογίζει σε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η παρουσίαση που ήθελα να σας κάνω εκ μέρους της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληρέστατη αυτή η παρουσίαση εκ μέρους της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ και θέλουμε να ακούσουμε και τι έχει να μας πει συνέχεια. Η κυρία Ρεγκογιάν Πέρες έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, βλέπω ότι έχουμε και πολύ καλή προσέγγιση όλοι οι σκιώδεις εισηγητές σε σχέση με αυτή την έκθεση και συμμερίζομαι και την ανάλυση κατά τα άλλα με την ανάλυση του κυρίου Ντεγιόν ακριβώς για την ανάλυση αυτού του θέματος υπό μια συνεκτική γραμμή, μια γραμμή που θα συμμερίζεται το έργο το οποίο αναπτύξαμε προηγούμενα και θα είμαστε συνεκτικοί με αυτό και με τον κοινό νου, την κοινή λογική για την αναζήτηση τη σωστή ισορροπίας μεταξύ μικρών καταστημάτων και μεγάλων καταστημάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κρίση που δημιουργεί η κρίση. Επίσης ε, και την δυνατότητα όσον αφορά την σωστή χρηματοδότηση και υποστήριξη. Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα και των ωραρίων εργασίας. Ξέρουμε πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να υπάρξει ανταγωνισμός σε σχέση με τέτοια ωράρια. Είμαι και εγώ υπέρ του να διασωθεί το λιανικό εμπόριο, να διασωθούν τα μικροκαταστήματα, διότι είμαι υπέρ της διοργάνωσης στις πόλεις μας με αυτά τα καταστήματα, στον κοινό χώρο που θέλουμε να αναπτύσσουμε με αυτόν τον τρόπο, στις γειτονιές ε, με τα μικρά καταστήματα. Έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα για τη ζωή μιας πόλης αυτό. Γι' αυτό η ανάλυση που απορρέει και οι προτάσεις που γίνονται από αυτή την έκθεση θα διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο την αναζήτηση αυτής της ισορροπίας, ώστε το λιανικό εμπόριο να μπορέσει να ενδυναμωθεί και να προαχθεί εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις δράσεις που προτείνονται στο πρόγραμμα δράσης. Είναι ικανοποίηση το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε κάποιες από τις ιδέες που εμφανίζονται στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο το 2011. Κυρίως σε αυτά τα οποία αφορούν τα σοβαρά προσκόμματα και εμπόδια όσον αφορά τα μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου, το λιανικό εμπόριο. Πρέπει να αρθούν αυτά τα προσκόμματα και τα εμπόδια στα θέματα των πληρωμών για παράδειγμα και των πρακτικών. Παρ' όλα αυτά θέλω να υπογραμμίσω ένα θέμα που για την ομάδα μου έχει προτεραιότητα. Πρόκειται για την πρόσβαση στην απασχόληση, την βελτίωση των όρων απασχόλησης και φυσικά την καταπολέμηση της παραοικονομίας στο λιανικό εμπόριο αληθεύει και το ξέρουμε όλοι ότι το λιανικό εμπόριο μπορεί να προαγάγει την πρόσβαση στην απασχόληση των νέων ή των μακροχρόνια άνεργων που θέλουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Πιστεύω και ότι είναι σημαντικό ότι αν στοιχηματίσουμε για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα αυτό πρέπει να επενδύσουμε επίσης στις δεξιότητες και ικανότητες και τα προτερήματα αυτών των εργαζομένων στην κατάρτισή τους. Οι δημοσιονομικές περικοπές στην κατάρτιση και την εκπαίδευση είναι αποτυχία και οπισθοδρόμηση διότι έχουμε απώλεια και μείωση του, απομείωση του ανθρώπινου δυναμικού συρρήκνωσή του. Θέλω να τονίσω την ε, ανάγκη να καταπολεμήσουμε την παράτυπη οικονομία, την ε, παραοικονομία και την εισφοροδιαφυγή. Πρέπει η εργασιακή νομοθεσία να εφαρμόζεται σωστά. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόταση του κυρίου Κορνέλης Ντε που είμαι σίγουρη ότι θα μας προσφέρει μια εξαιρετική βάση εργασίας για την προαγωγή μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς για το λιανικό εμπόριο που θα σέβεται τα δικαιώματα καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Λίκεργαρντ, ο κ. Μάντερς, η κυρία Ρούλα. Θα μιλήσω μετά εγώ και μετά η κυρία Στάιλερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Κ. Στεκάμπος μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Λούκεγκάρ. Δυστυχώ δεν είναι στις Βρυξέλλες και θα ήθελα να σας πω αυτά που ήθελε να θέσει. Λέει ότι είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ότι η Επιτροπή μας δίνουν σημασία ε, στο λιανικό εμπόριο, στον τομέα αυτό. Οι 11 προτινόμενες δράσεις είναι καλές. Το πρόβλημα συχνά είναι η επικουρικότητα, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά σε αυτόν τον τομέα Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις ευρωπαϊκές όσον αφορά το λιανικό εμπόριο που δυσκολεύουν τους ε, ανεξάρτητες, ε, τα ανεξάρτητα μαγαζιά να επιβιώσουν σε σχέση με τα μεγάλα καταστήματα και με μεγάλες αλυσίδες. Οπότε ε, είναι ομοιόμορφη επιλογή των καταστημάτων αυτόν τον τρόπο. Βλέπεις τα ίδια μαγαζιά παντού. Στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Βερολίνο κλπ και νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με τους κανονισμούς που προανέφερα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Είναι κάτι ε, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω συντονισμού μεταξύ των φορολογικών αρχών της Ευρώπης. Το σημαντικότερο δεν έχει αναφερθεί όμως. Ο ρόλος που παίζει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής αποφασίζει πού πάει να αγοράσει. Και ίσως λόγω των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας, της νέας τεχνολογίας, κινητών, τηλεφώνων, έξυπνων τηλεφώνων, τηλεόρασης κλπ. Ο καταναλωτής είναι αυτός που αποφασίζει τι και πού θέλει να το αγοράσει. Και εμείς ε, αποφασίζουμε να σώσουμε τα μικρά καταστήματα. Εγώ ζω σε ένα χωριό με 1.800 κατοίκους. Έχουμε ε, τον παπουτσί, έχουμε τον φούρναρι, όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα και το μικρό μαγαζάκι της γωνίας δύσκολα επιβιώνει. Διότι ο κόσμος παίρνει το αυτοκίνητό του και φεύγει και πάει στο σούπερ μάρκετ στη μεγάλη πόλη. Και πάει στο μαγαζάκι για να πάρει λίγο μαϊντανό αν το ξέχασε. Ο καταναλωτής δεν θέλει αυτά τα μικρά καταστήματα πια, ίσως. Ίσως μια λύση θα ήταν να το συμπεριλάβουμε αυτό στο πρόγραμμα, σχολικό πρόγραμμα των παιδιών. Να εξηγήσουμε στα παιδιά που θα είναι οι μελλοντικοί καταναλωτές ποια είναι η αξία των μικρών καταστημάτων και του λιανικού εμπορίου. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν μόνο στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Εκεί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Δεν έχω άλλες λύσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας για το θέμα και ελπίζω ότι τελικά ο εισηγητής θα ακολουθήσει μια πραγματιστική προσέγγιση στο πρόβλημα. Η κυρία Ρούλε. Χαίρομαι Γι' αυτό πολλά ενδιαφέροντα πράγματα αναφέρθηκαν. Θέλω να προσθέσω και εγώ τη φωνή μου σε αυτά που από πλευρά τη κοιόδου εισηγήτρια του ΕΛΚΑ αναφέρθηκαν. Πρέπει να βασιστούμε φυσικά στο σύνολο των προτάσεων που έχει εκπονήσει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και να μην επινοήσουμε τον τροχό εκ νέου από μηδενικού σημείου. Πολλά αναλύθηκαν τότε, διαπιστώθηκαν και ε, αυτό το οποίο βλέπω ότι κάποιε ελλείψεις έχει και θέλω να συμπληρώσω το είδαμε σε σχέση με τα θέματα της έκθεσης της κυρίας Κοράτσα Μπίλ. Το ότι λιανικό εμπόριο φυσικά διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην αποδοτικότητα της ενέργειας και την διαφύλαξη των πόρων και την ε, διασφάλιση των πόρων. Και τα απόβλητα και όλα αυτά διαδραματίζουν ένα ρόλο. Αρκετά έχουμε πετύχει και το φόρουμ θα πρέπει να εξετάσει ακόμα περισσότερο αυτή την πτυχή, αυτή τη συνιστόσα, διότι στην ενεργειακή αποδοτικότητα πολλά μπορούμε να πετύχουμε αν είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι το μόνο που θέλω να αναφέρω επιπρόσθετα στις παρατηρήσεις για το θέμα της διασφάλισης θέσεων απασχόλησης και σε σχέση με όσα είπε ο κύριος De Jong. Έχει δίκιο ο κύριος De Jong. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία μέσω κανονιστικών και ρυθμιστικών ρυθμίσεων μπορούμε να πετύχουμε πετύχουμε. Πολλά μπορούν να επιτευχθούν με βάση εθελούσε εθελοντικέ συμφωνίε. Διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε με τα μικρά καταστήματα στου χώρου τη Υπέθρου, στην Ήπεθρο. Είναι περισσότερο οι, οι ηλικιωμένοι οι οποίοι υποφέρουν από μια τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ αργά όταν δεν υπάρχει πια κάποιο ε, στην οικογένεια και τα καταστήματα αυτά κλείνουν κιόλα. Υπάρχουν ιδέε που είναι σωστέ από την άλλη όμως πλευρά. Δεν πιστεύω ότι με αυτή την έκθεση θα μπορέσουμε τόσο πολύ να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα και ώστε να καταφέρουμε να είμαστε πια, ας το πω έτσι, ε, ρηξικέλευτοι. Υπάρχουν πολλές μελέτες, πολλές αναλύσεις, είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτήσουμε αυτή την πορεία. Ευχαριστώ. Ε, Ίσως να κάνω κανένα δύο σχόλια κι εγώ. Νομίζω ότι ο Ντένις έθεσε διάφορα ζητήματα. Σωστά. Θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία η δουλειά τη Επιτροπή που διεξήχθη. Περιέχονται νέα στοιχεία, κάποια νέα στοιχεία. Πολλά αναφέρονται στην αλυσίδα των τροφίμων που είναι δική μα αρμοδιότητα, παρόλο που μα ενδιαφέρουν οι πτυχέ ε, που σχετίζονται τον καταναλωτή για αυτόν τον τομέα. Θα ήταν ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις ε, για τον εφοδιασμό στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ε, αν πλησιάσαμε σε, θελοντική, πλησιάσαμε σε θελοντική συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε. Κάποιε χώρε συμπεριλαμβανομένε τη δική μα εισάγουν αυτά τα μέτρα. Άρα έχουμε δημοσιολαβητή για την αισθήτα τροφίμων που υπάρχει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα έπρεπε να δούμε και τι βέλτιστε πρακτικέ και δραστηριότητε, λαμβάνοντα υπόψη βέβαια ότι σε κάποιου τομεί δεν έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά τι σχέσει επιχείρηση με επιχείρηση. Το ξέρουμε και στην οδηγία για τι της εμπορικέ πρακτικέ τι γίνεται και διάφορε πτυχέ που εξετάζει ο Ντένι για την παραπλανητική διαφήμιση. Που βεβαίω και αυτό μπορούσε να ισχύσει. Εδώ. Κάποιες σημαντικές πτυχές θα σχετίζονται με την πρόσβαση στην αγορά. Πολλή δουλειά που έκανε η Επιτροπή κυρίως στην πολιτική ανταγωνισμού, το επιλεκτικό τα φρέμ, τα πλαίσια ε, επιλεκτική διανομή όσον αφορά τι γνωστέ μάρκε. Είναι και αυτά σημαντικά. Κυρίω όσον αφορά τα μικρότερα καταστήματα που ίσω να ειδικεύονται για συγκεκριμένη μάρκα ε, προϊόντων που διαθέτουν. Και πόσο αυτά τα αγαθά είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο. Και πολλαπλή, πολλαπλής εφοδιασμός και διασυνοριακό εφοδιασμός είναι ένα άλλο ζήτημα. Επί ασχολιόμουν με τη διανομή των αυτοκινήτων και ήξερα ότι αυτό ήταν θέμα το δεκαετία του 80 και του 90 και η κυρία Ρέμπεν το έχει εξετάσει το θέμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ίσως εκεί μπορούμε να αντλήσουμε κάποια σημαντικά μαθήματα. Εκεί κοιτάζαμε και την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ των πολιτών, των αντιπροσώπων αυτοκινήτων και των προμηθευτών μάλλον λιανοπολιτών και των διανομέων ε, και ποιε ήταν οι πολιτικοί ε, όσον αφορά την τιμολόγηση, η πρόσβαση στα ανταλλακτικά κλπ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο λιανικό εμπόριο και αυτά. Και άλλα ζητήματα που ήδη επεξεργάζεται. Κόστος παραχή ε, παραρχής εφοδιασμού που το εξετάζει η αρμόδια γενική διεύθυνση και άλλε συναφείς πτυχέ. Ήδη κάποια από αυτά εκαλύφθησαν από την έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ και πρέπει να εξεταστούν εκ νέου. Η κυρία Ρούλε σωστά τα είπε αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα και την ετικετοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους πέντε βασικούς φορείς για πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες και βιώσιμες υπηρεσίες έβαλε την ε, ισχύ, την ε, επιρροή που είχε καταναλωτής. Αυτό που να το προσέξουμε ιδίω, κυρίως το πρόγραμμα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ε, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε όλες ιδιαίτερως ως αρμόδια επιτροπή για την προστασία του καταναλωτού αυτή τη φράση που λέει να δίνουμε εξουσία δύναμη στον καταναλωτή. Ε, παράλληλα πρέπει να σκεφτούμε και τη διάδραση μεταξύ διαθεσιμότητας online ε, διανομής δυναμικού υπάρχει εκεί με το τι προσφέρει η αγορά μπορεί να ξεκινά από φοδιασμό μικρού λιανοπολιτή μέχρι μια παγκόσμια αγορά και γίνονται πολλές μελέτες για ειδικού ε, ε, λιανοπολιτές που μεγάλωσαν, αναπτύχθηκαν και έφυγαν από το μικρό τους κατάστημα διότι πέρασαν από τη δύναμη που δίνει το διαδίκτυο γιατί τα προϊόντα τους είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο Ντένις ε, αναφέρθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τους μικρούς λιανοπολιτές. Δεν πρόκειται, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, είναι κάτι που απαγορεύει τους μικρούς λιανοπολιτές να μεγαλώσουν. Αυτό δεν μας πειράζει. Το μικρό μέγεθος δεν είναι το χαρακτηριστικό που ψάχνουμε, το εγενές, αλλά η ποιότητα της προσφοράς και η επιλογή που προσφέρεται. Είναι η ισορροπία. Μεταξύ αυτών προσφέρουν μεγάλα, τα μεγάλα καταστήματα και τα μικρά. Θέλουμε ένα χώρο που να μπορεί να μπει και ο λιανοπολιτής και να πουλήσει το ειδικό του προϊόν στο χώρο όπου πηγαίνουν άνθρωποι στο μεγάλο καταναλωτή. Δηλαδή παίζει ρόλο η κυκλοφορία των ε, καταναλωτών από ένα χώρο. Είναι περίπλοκο το κράμα. Δεν, είναι ένα, δεν μπορούμε να πούμε θέλουμε πολλά μικρά ε, μαγαζιά. Είναι ο συνδυασμό της προσφοράς στον καταναλωτή. Το, το, το, κράμα, το μείγμα, αυτό εξετάζουμε. Έχουμε ενδιαφέρουσα πρόκληση, ίσως να μην συμφωνούμε με όλα, αλλά με τα χαρά να συμμετάσχω στη συζήτηση, με ενδιαφέρει. Η κυρία Στάιλερ ε, θέλει και εκείνη να μας πει κάτι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και άλλους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω η περιπλοκότητα που αναφέρεται. Προερχόμαστε και από διαφορετικούς πολιτισμούς πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτά και κάποιες άλλες πτυχές. Μια άλλη πτυχή που μόνο ακροθυγός αναφέρθηκε είναι πώς θα ενθαρρύνουμε εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν μια τέτοια πρωτοβουλία στο ελληνικό εμπόριο για να μπορέσουν να βρουν μια τέτοια δυνατότητα το να συμμεριστούμε τις βέλτιστες πρακτικές είναι μια δυνατότητα. Για να υπάρχει η δυνατότητα να ανάληψεις μιας πρωτοβουλίας, να ξεκινήσει για παράδειγμα μια τέτοια δυνατότητα ε, για το 2013 ανοίγει μια τέτοια δυνατότητα με καινοτόμες δράσεις ε, για τον ανταγωνισμό και οι όσοι ε, κατέληξαν σε, ε, στην επιλογή και ε, επελέγησαν με ε, την βράβευση με τη δυνατότητα να ξεκινήσουν αυτά τα μαγαζιά και να ανταγωνιστούν για αυτή την περίοδο, δοκιμαστική περίοδο και θα υπάρχει η δυνατότητα απονομής αυτών των βραβείων 10.000 λιρών. Είναι η δυνατότητα να δοκιμαστεί αυτή η πρωτοβουλία με πρακτικό τρόπο οποιοδήποτε ξεκινά και στη δική μας ε, περιφέρεια και στο Ηνωμένο Βασίλειο όποιος θέλει να συμμετάσχει οι 10 αυτοί οι νικητές οι 10 που επελέγησαν για την ε, τελική αυτή δοκιμασία και άλλες δυνατότητες πρέπει να υπάρχουν από πλευράς άλλων κοινοτήτων για την ε, προαγωγή τέτοιων πρωτοβουλειών να μπορούν τέτοιες δυνατότητες να δοκιμαστούν πρακτικά και να προαθούν ώστε να μπορέσουμε με αυτού του είδους ε, τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών να προχωρήσουμε. Είναι καινοτόμα δράση. Είναι ο πολλαπλασιαστής ε, που έχει, ως, ε, έχει χαρακτήρα πολλαπλασιαστή αυτή η δυνατότητα. Αν δοκιμαστούν όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στην πρακτική εφαρμογή αυτών κατά το 2013. Μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα αυτή που ακολουθείται από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε, να υπαγάγουμε σε αυτές τις δυνατότητες όταν θέλουμε να ενισχύσουμε το λιανικό εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Πρακτικό και ενδιαφέρον παράδειγμα. Σίγουρα θα μας πείτε τα αποτελέσματα αυτών, ακόμα και αν δεν μπορούμε να έρθουμε την ίδια μέρα στον Τον Φέρμιν. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Ο Αντώνιο. Σε ευχαριστώ Μάλκομ. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Όλα οδηγούν στην στην αποσυναρμολόγηση, στην αποξύλωση των ε, μικρών ε, καταστημάτων λιανικού εμπορίου στις πόλεις μας, ε, το σύστημα φορολόγησης που διευκολύνει την φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή σε χώρες που δίνουν δυνατότητες σε τέτοιες δράσεις. Στην χώρα μου, για παράδειγμα, η μεταξύ εκείνων των χωρών που ε, και στις ε, ε, στα χρηματιστήρια βλέπουμε ότι πάρα πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ολλανδία διότι αποκομίζουν φορολογικά ωφέλη από μια τέτοια καταχώρησή τους εκεί Φυσικά όμως ε, υπάρχει και ο πολιτισμός στις χώρες μας, ε, για παράδειγμα, της καθημερινής επίσκεψης ε, σε τέτοια μικροκαταστήματα. Όμως η τάση βαίνει κατά αυτών των μικρών καταστημάτων. Οι εξελίξεις αντιβαίνουν αυτή την διατήρηση των μικρών καταστημάτων. Πρέπει λοιπόν να, ανατραπούν, να ανατρέψουμε τις τάσεις και να έχουμε και προγράμματα για την, ε, τον εξυγχρονισμό και την επικαιροποίηση σε ε, μικρή κλίμακα. Ωστόσο για την αγορά, για παράδειγμα, ε, εξοπλισμού ή για την ε, δυνατότητα να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε έστω την βιτρίνα ενός μαγαζιού. Αυτά δεν επαρκούν όμως. Χρειάζονται έντονες προσπάθειες συντονισμού και στον τομέα των περιφερειακών ταμείων και κονδυλίων για την προστασία καταναλωτών για παράδειγμα και υπό τους όρους ε, της φορολόγησης. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο εναρμονισμό, φορολογικό εναρμονισμό, αλλά συντονισμό ή δικαιοσύνη φορολογική που θα έπρεπε να προαγάγουμε. Κάθε μικρή προσπάθεια που μπορούμε να προχωρήσουμε και να προαγάγουμε θα ήταν θετική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονης ανεργίας. Για κάθε μικρό κατάστημα που κλείνει υπάρχουν τρία επιπλέον μέλη τρία άτομα που ε, θα καταστούν άνεργα. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά εδώ να δούμε τις ε, ε, εισφορές και τα επιδόματα ανεργίας που θα πρέπει να πληρώνονται και το τι συνεπάγεται αυτό υπό όρους κοινωνικής ασφάλισης και την απώλεια για παράδειγμα όσον αφορά ΦΠΑ και τα μισθώματα είναι μια καθαρή απώλεια λοιπόν όταν κλείνουν τέτοια μικρά καταστήματα. Δεν το εξετάζουμε παρκώς, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο. Ευχαριστώ. Good. I'm going to invite... Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέπνιντερ μήπως θέλει να πάρει το λόγο για να σχολιάσει αυτά που άκουσε ως τώρα και να μας πει οτιδήποτε άλλο θέλει βεβαίως. Και μετά ο κύριος ε, Μάντερς ε, να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλα τα ενδιαφέροντα σχόλια. Ε, χαιρόμαστε βέβαια όλος ιδιαίτερος που το πρόγραμμα δράσης μας για το λιανικό εμπόριο το βλέπετε θετικά. Και εμείς βεβαίως το βλέπουμε ως ε, συνέχιση μιας ε, διαδικασίας ε, που ξεκίνησε στην Επιτροπή σας και την οποία υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά το οποίο δείχνει τη σημασία του λιανικού τομέα και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ βεβαίως ήταν κρίσιμη σημασίας στη δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Επικροτώ λοιπόν την προσέγγιση αυτή και μπορεί να, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε είναι η μελλοντική μας συνεργασία. Βεβαίω θα, παρουσια... παρακολουθήσουμε το... τη στρογγυλή τράπεζα για το λιανικό εμπόριο με πολύ ενδιαφέρον, όπως επίσης και στο πλαίσιο μιας ε, ομάδας εργασίας ε, που εμείς θέλουμε να ε, οργανώσουμε στο πλαίσιο αυτής. Μάλιστα υπήρξε και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σήμερα ώστε να υπάρχει αυτό το αντανακλαστικό της Επιτροπής της, του Λιανικού Εμπορίου σε, στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις πολιτικές. Ε, μιλήσατε για ενημέρωση των ε, πολιτικών, ε, της πολιτικής προς τους καταναλωτές σε σχέση με τα όσα γίνονται στο λιανικό εμπόριο. Βέβαια αυτό πρέπει να συμβαίνει με κάθε πολιτική. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη συζήτηση για τα μικρά καταστήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τι είδους νέες νέα μικρά καταστήματα ε, μπορούν να ε, αναπτυχθούν. Δεν μπορώ να σχολιάσω όλα όσα ακούστηκαν σε αυτή την ε, πλούσια συζήτηση. Τα έχω, συζήτηση, τα έχω βέβαια σημειώσει όλα και θα τα λάβουμε υπόψη. Και θα τα συμπεριλάβουμε στις διαδικασίες από τη δική μας πλευρά. Όπως είπα θα υπάρξει αυτή η ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρακολουθεί το σχέδιο για το λιανικό εμπόριο και θα δούμε βέβαια κατά πόσο υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον ε, τα σχόλια για τις ε, θελοντικές ε, πρωτοβουλίες και το πόσο σημαντικό το θεωρείται αυτό, ακόμα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, πρακτικές θεμητές εμπορικές πρακτικές. Προσπαθούμε τώρα να συνοψίσουμε τη διαβούλευση που είχαμε για ε, το, την πράσινη βίβλο για το θέμα αυτό. Ε, πάνω από 200 απαντήσεις λάβαμε και για το τομέα το διατροφικό αλλά και για τους ε, υπόλοιπους ε, τομείς που αναφέρατε κι εσείς. Τώρα προβληματιζόμαστε δεν ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε με τα στοιχεία αυτά, γιατί έχουμε και μία εκτίμηση ε, επιπτώσεων για το θέμα αυτό και πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τις συζητήσεις στη δική σας Επιτροπή για τις πτυχές αυτές. Χαίρομαι που άκουσα ότι υπάρχει υποστήριξη για την εθελοντική πρωτοβουλία, γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υποστηρίζει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε βέβαια ότι έχουμε αυτήν την ε, διτή προσέγγιση, παράλληλα έχουμε και την ε, μελέτη αντικτύπου για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συμπληρώσουμε με κάποιο τρόπο την θελοντική πρωτοβουλία. Με χαροποίησε ε, το σχόλιο για την προσέγγιση ε, του καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής ε, είναι συχνά, πρωτοστατεί συχνά στο τι συμβαίνει στο λιανικό εμπόριο και αυτό βέβαια δεν είναι δυνατόν να μας διαφύγει όταν κάνουμε την ενημέρωση. Είναι δυνατόν να σχολιάσω όλες αυτές τις καλές ιδέες που άκουσα. Μόνο κάποια σχόλια μπορώ να κάνω. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι προσπαθούμε να εξελίξουμε κάτι ε, στο οποίο συνεισέφερε πάρα πολύ η Επιτροπή σας και ελπίζω ότι όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεργαστούν ώστε να ενημερωθεί αυτή η πολιτική. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να διατηρηθεί αυτή η ροή πληροφοριών. Και να αφορά τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, όταν θα ετοιμάσετε για κάποιο σχετικό έγγραφο, θα μας βοηθήσει. Θα δώσω το λόγο στον Ντένις Δε Γιόγκ για να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να μας ενημερώσει επί του χρονοδιαγράμματος. Ο Ντένις. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρες οι προτάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη. Βιωσιμότητα, απασχόληση, πτυχές καταναλωτού. Δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να διαφωνώ. Είναι πάντα θέμα ισορροπίας. και το να κεντρήσουμε το κείμενο σωστά πλαίσια. Θα είναι εφικτό. Το χρονοδιάγραμμα. Ξεκολουθεί να είναι το ίδιο το γνωστό. Σχέδιο έκθεσης θα πάει μέχρι 10 Ιουλίου για μετάφραση. Συζήτηση για δύο εκθέσεως 5 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία για τροπολογίες 10 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Έτσι λέει εδώ. Συζήτηση τροπολογιών 25 Σεπτεμβρίου. Εξέταση συμβαστικών τροπολογιών, κάτι καινούριο, κατόπιν αιτήματο της ΕΜΠΟ να καθυστερήσουμε κάπως. 17 Οκτωβρίου, έγκριση στην Επιτροπή 5 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, αντί του Νοεμβρίου. Διότι ΕΜΠΟ θέλει να ετοιμάσει σχέδιο γνωμοδότηση ΙΜΚΟ ε, και είναι καλό ε, να λαμβάνετε υπόψη το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής. Είναι καλό το ότι η Επιτροπή Απασχόλησης αναφέρεται συγκεκριμένα. Ίσως και η Επιτροπή Γεωργίας να μπει στον πειρασμό. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά είναι πολύ άσχολη αυτή. Πάντα. Θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσους, όσους πήραν το λόγο. Πάμε σε άλλη έκθεση νομοθετική, νομοθετικού περιεχομένου, πρόταση για οδηγία για προβασιμότητα των ιστοσελίδων των δημοσίων φορέων. Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης είναι ο εισηγητής μας που είναι παρόν. Έχουμε ολόκληρη ομάδα σκιωδών εισηγητών. Και ο Τσασκόφσκι, και ο Γκάς Βαρμόν, Έγκστρομ, ο κ. Μπίλαν απουσιάζει αλλά και εγώ μπορώ να πω μερικά πράγματα. Θα δώσω παρευθύ το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη για να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθέσεώς του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να αναφερθώ στη σημασία του ζητήματος πλέον. Ήδη έχει γίνει αυτό επανειλημμένα στην Επιτροπή. Οπότε θα πάω κατευθείαν στα αποτελέσματα της συνεδριάσεως των Σκιαδών της 14 Μαΐου και όλα τα ονόματα που αναφέρατε πρόεδρε ήταν άνθρωποι που ήταν παρόντες και ευχαριστώ όλους οι ιδιαίτερους για την άριστη συνεργασία η οποία οδήγησε άμεσα στο αποτέλεσμα το οποίο θα σας παρουσιάσω εδώ. Έλαβα έξοχη συνδρομή από τους συναδέλφους, προσπάθησα να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου τις προτάσεις και όλοι συμφωνήσαμε καταρχάς ότι η νομοθεσία εσωτερική αγοράς αποτελεί τη νομική βάση. Αυτή είναι η αφετηρία θα εστιαστώ στην παρουσίασή μου επί πέντε σημείων. Πρώτα απ' όλα το πεδίο εφαρμογή, μετά εποπτεία και υποχρέωση ενημέρωση και υποβολή αναφορών από τα κατημέλη, κυρώσει, το τρίτο στοιχείο. Αναθεώρηση οδηγία μετά είναι το τέταρτο. Και στο τέλος θα αναφερθώ στους ορισμού. Θα ξεκινήσω με το πεδίο εφαρμογή. Όλοι πιστεύαμε ότι το πεδίο εφαρμογής που είχε επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ περιορισμένο, πολύ στενό και οι περιορισμένε αυτέ οι υπηρεσίε, ε, ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σωστό, δεν πετυχαίνει το σκοπό. Διευρύναμε λοιπόν το πεδίο εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα και του φορεί και στι σελίδε των φορέων αυτών των δημοσίων για να πετύχουμε σταδιακή εφαρμογή των μέτρων μέχρι το 2020, για να επιτρέψουμε την επίτευξη των στόχων σε εύλογο χρονικό διάστημα, εισάγαμε ένα νέο μοντέλο φορμογής, όπου οι ιστοσελίδες των δημοσίων φορέων λειτουργούν σε εθνικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτοί που είναι σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα, θα λειτουργούν στο 2016, σε περιφερειακό 2018 και σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2020. Αυτά είναι τα όρια. Ε, ξέρω ότι η βασική αντίσταση προέβη από την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτή καλύπτεται. Έχει περισσότερο χρόνο η τοπική αυτοδιοίκηση με αυτή την πρόταση. Αλλάξαμε κάπως την όλη φιλοσοφία και χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πετύχαμε αυτό που μας βοήθησε να βρούμε τη λύση. Νομίζω ότι είναι άριστη η λύση διότι σε πολλές χώρες δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ εθνικού ή ομοσπονδιακού επίπεδου και περιφερειακού. Γι' αυτό ε, θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιστοσελίδων με την μετατροπή των εθνικών ιστοσελίδων ήδη θα καλύπτεται. Με την έκθεση προχωρώ και ένα βήμα πιο πέρα και στα παραρτήματα. Στο παράρτημα βάζω και έναν κατάλογο των βασικών υπηρεσιών προς το κοινό που προσφέρονται από ιδιωτικούς φορείς. Ήταν μεγάλη συζήτηση αυτή πώς να αντιμετωπίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται από τους ιδιωτικούς φορείς. Και μέχρι το 2020 και οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να, καλύπτουν τις κάτωθοι υπηρεσίες, ε, ηλεκτρικές, ενέργεια, αέριο, ε, ταχυδρομικές ε, υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και υπηρεσίες, τραπεζικές, ασφαλιστικές υπηρεσίες, πρωτογενής, δευτερογενή, υψηλή, τροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, συμπληρωματική ασφάλιση, υγειονομικές υπηρεσίες και περίθαλψη των παιδιών, παιδική μέρημνα για τα παιδιά και έχουμε μια εξαίρεση στην οδηγία που είναι οι μικροεπιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ 10 εργαζομένους. Μέχρι το 2020 όλες οι σελίδες που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και που καλύπτονται θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από το κοινό. Αυτό αντικατοπτρίζει και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ανθρώπων με ε, αναπηρίες και έχουμε μείνει πίσω σαν Ευρωπαίοι και έτσι θα ευθυγραμμιστούμε και με τις διεθνείς υποχρεώσεις που υπέχουμε. Θα στραφώ τώρα προς το δεύτερο τμήμα της παρουσιάσεως, εποπτεία, έλεγχος και υποβολή αναφορών. Αυτή ήταν μια άλλη έλλειψη που εντοπίστηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ ήταν λογικό να χωρίσουμε τα ζητήματα εποπτεία και υποβολή αναφορών και να εισάγουμε δύο ξεχωριστά άρθρα για τα θέματα αυτά. Έτσι η οδηγία γίνεται πιο ευανάγνωστη και περιγράφονται και οι δύο υποχρεώσει. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα με την εποπτεία και τον έλεγχο. Τα κράτη-μέλη θα καθορίζουν καταρχά αρμόδιε αρχέ, την αρμόδια αρχή που θα ελέγχει την εφαρμογή τη οδηγία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αρχή τη επικουρικότητα η καθοριστής αρμόδια αρχή και το κάτω μέλος μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα ποια αρχή θα επιλεγεί επίσης θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση εδήποτε καταγγελιών που θα υποβάλλονται από χρήστε ή ενδιαφερόμενα μέρη εσδήποτε αποτυχίες συμμόρφωσης όσον αφορά τις απαιτήσει για προσβασιμότητα σε λόγω ιστοσελίδες. Είναι σημαντικός ο μηχανισμός για την υποβολή καταγγελιών, διότι οι πολίτες με αναπηρίες που είναι βασικό στόχο της οδηγίας θα μπορούν να καταγγέλουν προβλήματα με προσβασιμότητα, την έλλειψη προσβασιμότητας κάποιες τοσελίδες Είναι ανοιχτή η διατύπωση και έχουν το δικαίωμα οι ίδιοι να απευθύνονται στι αρμόδιε αρχέ. Τα κάτι μελη θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να ενημερώνουν του χρήστε ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δυνατότητα κατάθεση καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή καθ' αυτή θα δημιουργήσει ομάδα εργασία που θα αποτελείται από εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπου που θα διορίζονται από τα κράτη-μέλη, που θα αντιπροσωπεύουν τι αρμόδιε αρχέ και θα συναντώνται τακτικά αυτοί κατόπιν προσκλήσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να συζητούν για τα αποτελέσματα του ελέγχου και για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλού τομεί. Δεν προβλέπεται στην οδηγία και το συμπεριλάβαμε σε αυτή την οδηγία. Και τώρα να αναφερθώ στην υποβολή αναφορά. Τακτικά τα κάτι μελη θα υποβάλουν αναφορέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Και είπαμε τακτικά, δεν είπαμε ετησίωση κάθε δύο χρόνια. Τακτικά, για να τα αφήσουμε ανοιχτό. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε γραφειοκρατικό άχθο. Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν το δικό του το ρυθμό, αλλά αυτή η έκθεση θα δημοσιοποιείται και θα έχει προσβάσιμη μορφή. Ανοιχτή μέθοδος λοιπόν που επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση στις εκθέσεις και εάν χρειαστεί να υποβάλω μια καταγγελία. Μετά στρέφομαι στο τρίτο τμήμα της παρουσιάσεώς μου, της κυρώσεις. Τα κράτη-μέλη, δεν προβλεπόταν αυτό έτσι, οι κυρώσει δεν προβλεπόταν μέχρι τώρα. Τα κράτη-μέλη θα καθορίζουν του κανόνε περί κυρώσεων, τα ίδια τα κράτη-μέλη, για κυρώσει που εφαρμόζονται και παραβιάσει των εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται δυνάμει τη οδηγία αυτή και θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτω ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι κυρώσει θα εφαρμόζονται. Είναι μια μέθοδο ε, η οποία βρίσκεται και σε άλλου τομεί τη ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Και τώρα να έρθω στο τέταρτο τμήμα, που είναι η αναθεώρηση τη ε, οδηγία είναι ένα νέο στοιχείο που εμείς σαν κοινοβούλιο θα θέλαμε να συμπληρωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβαίνει σε αναθεώρηση οδηγίας μετά από τρία χρόνια διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν μια αξιολόγηση, έκθεση αξιολογήσεων που θα υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να μπορεί να δει κατά πόσο οι στόχοι τη οδηγία έχουν επιτευχθεί από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να κλείσω με το πέμπτο κομμάτι, του ορισμού Σύμφωνα με το νέο πεδίο εφαρμογή που έχουμε εισάγει, προσθέσαμε και νέους ορισμούς. Δεν πρόκειται να διαβάσω τους ορισμούς. Θα ήθελα όμως να τονίσω ποιες βασικές λέξεις έχουμε καλύψει με ορισμούς. Πρώτα απ' όλα, προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα. Τι σημαίνει προσβασιμότητα. Μετά καθορίζουμε τον φορέα του δημόσιου τομέα μετά ορίζουμε τις ιστοσελίδες που ανήκουν στον φορέα του δημόσιου τομέα και οι ιστοσελίδες που παρέχονται από φορείς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους καταναλωτές. Είναι σαφείς οι διαχωρισμοί. Και έχουμε και ορισμό για, για τεχνολογία που βοηθά, που βοηθά. Είναι βασικό θέμα διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο στους σελίδες αλλά και κινητές συσκευές και κυρίως αμφίδρομη διάδραση, συμπλήρωση, ε, ταυτοποίηση, ε, πληρωμές, όλες αυτές οι διαδικασίες καλύπτονται. Ο ορισμός των καλυπτωμένων ιστοσελίδων και περιεχόμενων των ιστοσελίδων αναφέρονται σε αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα να αναφερθώ εκτενέστα σε αυτό. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, website concern, αναφέρεται σε όλες τις εκδοχές των σελίδων που καλύπτονται από την οδηγία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχω σχεδιαστεί για είναι προσβάσιμες μέσω κινητή συσκευή ή με άλλο μέσο. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσπαθούμε να μην δούμε μόνο τι γινόταν στο παρελθόν, αλλά το παρόν και λίγο ε, προς το μέλλον στρεφόμαστε. Η επικείμενη, ε, επόμενη Λιθουανική Προεδρία ευτυχώς την νομοθεσία αυτή την έχει βάλει στον κατάλογο προτεραιοτήτων και πιστεύουμε ότι η επόμενη Προεδρία που θα ξεκινήσει το 2014 και η Ελληνική Προεδρία θα ολοκληρώσει αυτή την νομοθεσία, η Ελληνική ε, Προεδρία. Λοιπόν, ας συνεργαστούμε για να ε, μειώσουμε τις φραγμούς που υπάρχουν στο διαδίκτυο για ανθρώπους ε, οι οποίοι πράγματι χρειάζονται μια άρση αυτών των εμπόδιων στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητής. Σκιώδης εισηγητές. Τσασκόφσκι. Πρώτος και καλύτερος. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά μόλις τελειώσω την παρέμβασή μου, πρέπει να τρέξω στην Αύκο γιατί συζητείται εκεί η έκθεσή μου. Πρώτον, να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή γιατί συνεργαστήκαμε πολύ και έχουμε την ίδια φιλοσοφία να είναι λίγο πιο φιλόδοξη αυτή η έκθεση. Συμφωνώ σχεδόν με όλες σας τις ανησυχίες και σχεδόν με όλες σας τις ιδέες ε, για την, ε, το να αλλάξουμε λιγάκι το ε, σχέδιο πρότασης της Επιτροπής. Πρώτον, όσον αφορά τους ορισμούς, γιατί όταν μιλάμε για, εθνικούς, για εθνικό, τοπικό, περιφερειακό, Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γερμανική ιδιαιτερότητα, αλλά αν σκεφτούμε τι προβλήματα έχουν ε, οι δημόσιοι φορείς ε, με την προσβασιμότητα, ε, είναι κυρίως ε, το εθνικό επίπεδο, είτε είναι εθνικό, είτε είναι ομοσπονδιακό, είτε σε επίπεδο κρατηδίων. Και μετά είναι και το τοπικό επίπεδο. Δηλαδή δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διάκριση μόνο. Εθνικό και τοπικό. Το εθνικό να καλύπτει και το ομοσπονδιακό και το του κρατηδίου, γιατί ουσιαστικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που έχει τα βασικά προβλήματα. Οπότε δεν καταλαβαίνω αν χρειάζονται αυτέ οι τρει κατηγορίε, μήπω θα ήταν καλύτερο να έχουμε δύο. Και αν έχουμε τρεις κατηγορίες είναι και το πώς θα τις οριοθετήσουμε. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε την ορολογία ΝΑΤΣ, θα χρησιμοποιήσουμε ε, του ΩΣΑ. Είναι καλύτερο να είμαστε ακριβείς. Αν έχουμε δύο κατηγορίες, νομίζω ότι είναι πολύ σαφές τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είναι αυτονόητο γιατί το, το, το, το τοπικό επίπεδο είναι σαφώς οριοθετημένο στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη. Ε, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θα, συμφων, θα συμφωνούσαν να συμπεριληφθούν ε, και ιστότοποι που χρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μιλάτε για τακτική εκπόνηση εκθέσεων, ε, regular reporting λέτε. Ίσως θα πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο ακριβές, κάθε δύο-τρία χρόνια, γιατί ενδεχομένως η ετήσια έκθεση ίσως να είναι πάρα πολύ βαρύ. Να είμαστε όμως παρόλα αυτά πιο ακριβή. Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις ε, και την εξαίρεση, την εξαίρεσή άρχισα να το σκέφτομαι και συμβουλεύτηκα και κάποιους από τη χώρα μου. Μπορεί να είναι προβληματικό κάτι τέτοιο, γιατί για παράδειγμα... Ο τομέας της υγείας μας και οι υπηρεσίες υγείας ε, υπάρχουν ε, πολλοί που θεωρούν ότι είναι πολύ, πολύ λίγες οι επιχειρήσεις ε, αυτοαπασχολούμενων και προσπαθούν να χωρίζουν κάπως τις συμβάσεις. Ε, ε, υπάρχει δηλαδή μια μεγαλύτερη εταιρεία η οποία είναι τέλος πάντων ε, διαιρεμένοι σε μικρότερες ε, εταιρείε. Δεν ξέρω, αντί να τις εξαιρέσουμε, μήπως ήταν καλύτερα να τους δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. 2020, για παράδειγμα, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι τι εννοούμε μικροεπιχειρήσεις. Αν είναι ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, που έτσι γίνονται οι συμβάσεις, στην Πολωνία τουλάχιστον έτσι γίνεται, ε, ίσως δεν θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Οπότε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς. Η αρχική μου εμένα αντίδραση θα ήταν να μην τους εξαιρέσουμε, αλλά να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο. Τέλος, ε, η εφαρμογή των ε, κινητών. Ήρθα σε επαφή, συμβουλεύτηκα κάποιους εμπειρογνώμονες, γιατί το πιο σημαντικό είναι να είναι στο δυνατόν σαφέστερος ορισμός. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν μιλούμε για mobile applications, όταν μιλάμε για ιστοτόπους οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι σε ε, κινητά και τα αποκαλούμε εφαρμογέ, εντάξει, καλό είναι. Ε, αλλά αν μιλάμε για εφαρμογές κινητού τηλεφώνου, είναι, είναι αυτές οι apps, οι εφαρμογές που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα, που είναι κάτι διαφορετικό. Και επειδή μίλησα με πυρογνώμονες, ε, χρησιμοποιεί, χρησιμοποιεί το ATAG, αυτή την προδιαγραφή. Οπότε είναι λίγο πιο προβληματικό. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς τι θέλουμε να πούμε. Αν εννοούμε ιστότοποι προσαρμοσμένοι σε κινητά, σε κινητά πρόσβαση από κινητά, ε, ή αν θέλουμε να μιλήσουμε για εφαρμογέ κινητού τηλεφώνου, που είναι κάτι διαφορετικό. Και αν θέλουμε αυτό να κάνουμε, το δεύτερο, τότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώ θα το κάνουμε, με τι προδιαγραφές, με το κατά πόσο αυτό διευρύνει το πεδίο εφαρμογή ε, τη οδηγία με τρόπο που να είναι αποδεκτό και, αποδεκτός κλπ. Ε, όπως βλέπετε λοιπόν, ε, είναι μικρά ε, πράγματα αυτά. Το μόνο σημαντικό είναι ε, η οριοθέτηση κρατικού, ε, εθνικού και τοπικού. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι πρέπει να τα δούμε για να, είμαστε, να, να μιλούμε περισσότερο επί της ουσίας. Συγγνώμη που φεύγω, αλλά θα είμαι σε επαφή με τις εργασίες σας. Το καταλαβαίνουμε, λέει ο κύριος Πρόεδρος. Έχετε ε, ε προβλήματα γιατί πρέπει να πάτε στην ε, επιτροπή στην οποία συζητιέται η έκθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ συγχαίροντας τον εισηγητή, τον κύριο Χατζη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, που θα μας διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το να σημειώσουμε πρόοδο και να κινηθούμε προς μια κοινή πρόταση με σημαντικό περιεχόμενο και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενος πρόταση. Στην συνάντηση που είχαμε ήδη εξέφρασα την άποψή μας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε επί της ουσίας της οδηγίας και στην διεύρυνση του περιεχομένου και για τις διορίες και προθεσμίες εφαρμογής και τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και έλεγχο. Σε αυτό το βαθμό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιοι οργανισμοί και φορείς δημόσιοι θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και υλοποίηση της οδηγίας και για την παρακολούθηση επίσης, ώστε να ευνοήσουμε την παρουσία των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και των ε, οργανώσεων που, που εκπροσωπούν τα άτομα αυτά και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε με άλλα λόγια όλη αυτή την παρακολούθηση και συνέχεια που χρειάζεται για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Τώρα όσον αφορά την έκθεση θα ήμουν υπέρμαχος του ότι θα πρέπει να έχουμε μια ετήσια έκθεση και αυτό επειδή τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση αυτό γιατί αυτή η οδηγία έχει μεγάλη εμβέλεια, μεγάλο εύρος και όχι, όσο περισσότερα κάνουμε ώστε στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα βήματα ε, να είναι πραγματική εφαρμογή αυτής της οδηγίας, τόσο το καλύτερο για το μέλλον. Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής τώρα, συμπίπτω και συμφωνώ με τον εισηγητή Χατζημαρκάκη για την αναγκαιότητα που υπάρχει, την ανάγκη να διευρύνουμε τον κατάλογο που εμφαίνεται και φυσικά και νέες σελίδες που πρέπει να ανοίξουν στην ιστοσελίδα που πρέπει να είναι προσπελάσιμες, προσβάσιμες ευθύς εξ αρχής για όλους αυτούς. Με τέτοιο τρόπο ώστε με αυτόν τον τρόπο για την εφαρμογή του καταλόγου να αναφέρεται στο παράρτημα τι θα συμβαίνει, ποιοι θα είναι αυτοί για να, είναι, να είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι και εύκαμπτοι. Όσον ε, αφορά τον τομέα τον κρατικό, τον ομοσπονδιακό, τον τοπικό, τον περιφερειακό, Νομίζω στους περιφερειακούς και κρατικούς τομείς είναι αρκετά σαφές σε όλες τις περιπτώσεις τι θα γίνεται. Στο τοπικό όμως επίπεδο θα πρέπει να εξετάσουμε και την δυνατότητα ενός ε, ε, ορισμού που θα αναφέρεται σε βάση με τον αριθμό κατοίκων όσον αφορά τις ιστοσελίδες. Όχι μόνο απλά και μόνο να έχουμε την, ε, την αναφορά για κάθε χώρα του τοπικού επίπεδου, ώστε όταν έχουμε πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εντάξουμε κάποιες προθεσμίες και διορίες εφαρμογής και υλοποίησης πιο γοργές, πιο σύντομες από ότι στο τοπικό επίπεδο με μικρότερο πληθυσμό από 100.000 κατοίκους. Τώρα για τις προθεσμίες θα ήμουν πιο φιλόδοξος από ότι ο εισηγητής εδώ για τις προθεσμίες ο εισηγητής κάνει λόγο για προθεσμίες μέχρι το 2018-2020. Είναι όμως πολύ μεγάλες προθεσμίες αυτές για τις απαιτήσει όσον αφορά την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Θα ήταν πιο πρακτικό, θα ήμουν πιο υπέρ του να μειώσουμε αυτές τις προθεσμίες. Ανάλογα με τα επίπεδα 2016, 2017 18 ως χρονικές προθεσμίες. Και τέλος, Επίσης συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή του προλαλήσαντα για την ανάγκη να αναζητήσουμε δυνατότητες χρήσιμες και ωφέλιμες για την κινητή τηλεφωνία και τις λύσεις που θα προτείνονται και τις καινοτόμες τεχνολογικές ε, ε, λύσεις που επιταχύνονται. Όλα αυτά πρέπει να αποσαφηνίζονται στην οδηγία πώς θα λειτουργήσουν. Σε σχέση με τον κατάλογο που θα αναφέρεται στα παρατήματα, συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή. Ίσως θα έπρεπε εδώ σε ένα μικρότερο επίπεδο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα σε σχέση με τη διαφοροποίηση που προτείνεται για την κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων όσον αφορά και τα σημεία για την ενημέρωση και τουρισμό που αυτή τη στιγμή ε, δεν καλύπτονται ή τουλάχιστον κέντρα πολιτισμικά που δεν, έχουν, δεν συμπεριλαμβάνονται. Με όλα αυτά θέλω να πω πρόεδρε ότι κρίνω, πιστεύω ότι θα υπάρξει πολύ ευρεία, ευρύτατη συνένεση στο τέλος και οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί θα καλύψουν και θα καθορίζουν καλύτερα ή θα βελτιώνουν κάποιους τομείς που έχει προτείνει ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Thank you very much for your... Uh, Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Έγκστρομ από τους Πράσινους. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά του. Όταν ε, το συζητούσαμε το θέμα ως τώρα, εγώ έλεγα πάντα ε, ότι η ιδέα της Επιτροπής να αρχίσουμε με ένα περιορισμένο αριθμό ιστοτόπων ε, για να υπάρχει αυτό το, αυτός ο αντίκτυπος μετάδοσης από το ένα στο άλλο, εγώ συμφωνώ με αυτό, αλλά στην αρχή συμφωνούσα, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη, ειδικότερα επειδή Μίλησα με την ε, Ένωση Τυφλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν τη δική τους εμπειρία και εκείνη. Έχουμε προσπαθήσει κάποια ήπια μέτρα να ακολουθήσουμε κατά τα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Στην Αμερική έχουν νομοθεσία συγκεκριμένη και λειτουργήσε. Οπότε λοιπόν, ε, ό,τι είπα σε σχέση με αυτό, διαγράψτε το, άλλαξε γνώμη. Χαίρομαι σε γενικές γραμμές πάρα πολύ με το σχέδιο της γνωμοδότησης που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. το βλέπω να προχωράει πολύ γρήγορα. Αν έχουμε τροπολογίες, ε, πιστεύω ότι θα αφορούν κυρίως λεπτομέρειες ε, και τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους κοιόδης εισηγητές ε, για την ώρα. Να δώσω τώρα το λόγο στον Ηλία Ιακωβίδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θέλετε να σχολιάσετε κι εσείς. Σημειώνω την πολύ μεγάλη φιλοδοξία που υπάρχει. Βλέπω ότι παρατηθήκατε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινηθείτε για τα πάντα. Να μην πιστέψετε τη στρατηγική με τον λάχιστο κατάλογο της ασημένιας σφαίρας, αλλά να καλύψετε όλες τις δημόσιες ιστοσελίδες σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο τουλάχιστον. Κάποιες χώρες πάει πιο κάτω, σε 23 από τις 27 χώρες μέλια. Αυτή ήταν δική μας λογική. Δεν την εμπιστευτήκατε. Μιλήσατε με τους διάφορους εθνικούς φορείς και έχετε πιο φιλόδοξο στόχο. Τελικά το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε στο μυαλό μας. Εμείς είχαμε πιο μινιμαλιστική προσέγγιση από σας. Αυτό για το πεδίο έχω να πω. Εμείς διαλέξαμε την ελάχιστη παρέμβαση, την ασημένια σφαίρα, όπως την αποκαλώ, που θα επηρεάζονται μέσω Εθνικών Κοινοβουλίων όλες οι δημόσιες ιστοσελίδες. Το θέμα είναι του ελέγχου μας προβλημάτισε αυτό. Δημιουργήσαμε τις ιστοσελίδες. Ε, και θα παρακολουθείτε συγκεκριμένο αριθμό από τις ιστοσελίδες. Το να βάζετε όλες τις δημόσιες σελίδες. Συν αυτές που προσθέτεται για τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο ελεγκτικός φορέας. Παρακολούθηση που θα βασίζεται σε καταγγελίες ή ενεργή παρακολούθηση και εποπτεία από τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά είναι ανέφικτο. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ιστοσελίδες. Από τις τροπολογίες δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα εφαρμοστεί ο έλεγχος ή η εποπτεία. Στην πρότασή μας έχουμε την εφαρμοστική πράξη. Θα είχαμε ορισμένο αριθμό ιστοσελίδων που θα ελέγχονται τακτικά. Δεν ξέρουμε τι θα πούν και τα κράτη-μέλη, αν μια φορά το χρόνο ή ποιο θα είναι το διάστημα του ελέγχου. Άρα συνδυαζόταν το πεδίο κάλυψης εφαρμογής με τον έλεγχο. Επρόσδεκτε οι άλλες ιδέες, κυρίως για τον κινητό τομέα, αλλά προσέξτε. Από τη στιγμή που θα Μην ξεφύγουμε από τις προδιαγραφές που θέλουμε να εφαρμόσουμε λόγω των ε, κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Θα, θα φύγουμε από τον κορμό της οδηγίας. Εσωτερική αγορά επί οριζόντιας προδιαγραφής. Οι εφαρμογές αυτές πηγαίνουν εκτός του πεδίου. Ναι, για αυτή την οδηγία, οι ιστοσελίδες και το περιεχόμενο που θα είναι ε, προσβάσιμο από τα κινητά, αλλά οι εφαρμογές των κινητών θα είναι εκτός τα apps. Αυτή είναι η δυσκολία που διαβλέπω όσον αφορά την πλευρά μας. όταν είσαστε πολύ φιλόδοξοι ξέρετε τι κάνετε και με τα κράτη-μέλη, ελπίζω. Δεν θέλω να κολλήσει το θέμα, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και κρατών μελών. Αγεφύρω το χάσμα. Και έτσι θα περάσουμε στην επόμενη θητεία και ίσως ε, θα μείνουμε πολλά χρόνια πίσω θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, ευελιξία για να βρεθεί μια λύση με τα κάτι μελη Τα περισσότερα σχόλια όμως ε, μας βρίσκουν συμφώνους και ο τελικός στόχος είναι ο ίδιος ο δικός μας. Λοιπόν, συναντήθηκα με τη Λιθουανική Προεδρία το πρωί και έχουν φόρτο εργασίας. Και καταλαβαίνω αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνετε, θέλετε να κάνετε εσείς ως εισηγητής. Να στείλετε ισχυρό πολιτικό μήνυμα και να παραμείνει αυτό για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου ή να προχωρήσει το θέμα τώρα. Ίσως χρειάζονται κάποιες συζητήσεις ή εσείς να συζητήσετε με την ε, Λιθουανική Προεδρία για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει το όλο θέμα. Από τις συζητήσεις επίστωσα ότι δεν θεωρούν ότι είναι προτεραιότητα αυτό το θέμα, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η ασφάλεια των πληροφοριών κλπ. Αυτά είναι πιο σημαντικά για αυτούς. Άρα πρέπει να τους πείσετε ότι είναι προτεραιότητα. Ε, το αφήνω στη δική σας δύναμη της πυθούς. Θέλετε να ολοκληρώσετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με ενθαρρύνετε να δώσω συνέχεια σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε μια κατάσταση εκβιασμού. Αν υπαρχουν κάτι κράτη-μέλη που λένε ότι αυτό θα ήταν δαπανηρό και ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και μας εκβιάζουν και λένε αν κάνετε αυτό θα υπάρξει αυτή η συνέπεια, θα αναβληθεί μέχρι την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, εμείς θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη και στα, στους πολίτες να το πούμε αυτό απροκάλυπτα. Γιατί αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι υπερφιλόδοξο. Κατανοώ και έχω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για όλα τα σχόλια των συναδέφων. Κατανοώ ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο περιθώριο για καλύτερο ορισμό. Τι εννοούμε με εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Και θα μπορούσαμε, αν τα κράτη-μέλη αισθάνονται ότι υπάρχει κίνδυνος από αυτή την πρόταση εις βάρος τους να συγχωνεύσουμε το περιφερειακό με το εθνικό και να πούμε το 2016 να γίνει αυτό. Αλλά αυτό ήδη είναι καθυστερεί κατά πολύ τα πράγματα για πολλούς. Τώρα, για τη διαπραγμάτευση θα μπορούσαμε ίσως να αναζητήσουμε ένα καλύτερο ορισμό, καλύτερους ορισμούς σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν ο κύριος Τσεσκόσκι, ο κύριος Ραμών όσον αφορά την ετήσια υποβολή εκθέσεων. Αλλά αυτό κατά τα άλλα είναι κάτι το οποίο επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη. Να μην υπάρχει δηλαδή ε, δεσμευτική υποχρέωση να υποβάλλονται τέτοιες, εκτίσεις, ε, τέτοιες εκθέσεις με αυτό το πλαίσιο. Τώρα, θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι δεν την κάνατε εσείς αυτή την πρόταση, αλλά οι άλλοι δύο συνάδελφοι την υπέβαλαν. Και αν υπάρχουν δυσκολίες τώρα σε σχέση με την νομοθεσία ε, από πλευράς της Επιτροπής, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό, π.χ. μετροπολογίες Γενικά όμως, καθότι γνωρίζω ότι έχει ενταχθεί στον πίνακα προτεραιοτήτων, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων της Λιθουανικής Προεδρίας, ευελπιστώ ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε στο τέλος τέλος τη δική σας υποστήριξη και βοήθεια, Μάκομ Χάρμπορ. Ένα πράγμα είναι η τοποθέτηση του εισηγητή, οι σκιώδεις εισηγητές πορεύουν προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά χρειαζόμαστε φυσικά και την βοήθεια και υποστήριξη του Προέδρου μας. Ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας λέει ο κύριος Μάκομ Χάμπορ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει για να αναφερθούμε στο χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες. Εκπνέει προθεσμία 30 Ιουλίου. Τροπολογίες θα εξεταστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα περάσουμε στην επόμενη Ολομέλη τον Νοέμβριο. Θα υπάρξει λοιπόν επαρκής χρόνος για να εξεταστούν όλα αυτά. Ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν υπερφορτωμένο απόγευμα όσον αφορά αυτό το πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες μας. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση σημαντικού αριθμού τροπολογιών σε σχέση με τη γνωμοδότηση της κυρίας Γκαλό εξ ονόματος Επιτροπής Βιομηχανίας και θα ήθελα να πω ότι έχουμε 311 τροπολογίες μαζί με τις δικές σας. Κάπως με εξέπληξε και εμένα αυτό το θέμα για την έκθεσή σας. Να δούμε τι θα καταφέρουμε να κάνουμε. Πόσους και εισηγητές έχουμε για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Δεν παρίσταται η κυρία Πρέντεγκαστ. Ο κύριος Μπούσο, εσείς αναλαμβάνετε. Εντάξει ο κύριος Χατζημακάκης και αυτόν, ο κύριος Έγκστρομ και εγώ είμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν θα αναλάβουμε εμείς αυτό το θέμα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Κυρία Γκαλό, ποιες είναι οι απόψεις σας για αυτές τις τροπολογίες και κατά τα άλλα. Έχουμε και τον Άντρα Σέβιντα, τον καλωσορίζουμε που τακτικά παρακολουθεί τις ε, συναντήσεις μας. Να μας δώσει επίσης να ακούσουμε και την άποψη της Επιτροπής. Έχετε τον λόγο Μαρία Γκαλό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι, όπως και εσείς, λόγω του αριθμού των κατατεθισών τροπολογιών για το σχέδιο κανονισμού που αφορά την ταυτοποίηση την ηλεκτρονική και τις ε, υπηρεσίες ε, πιστευτικού χαρακτήρα στο online. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το θέμα, κυρίως μετά από μια πρώτη ανάγνωση των τροπολογιών είδα ότι υπάρχει κοινή θέληση να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ε, στον ψηφιακό τομέα. Θα προβώ σε μια παρατήρηση. Οι συνάδελφοί μου δεν ήταν όσο σχολαστικοί όσο και εγώ όσον αφορά το σεβασμό του άρθρου 50 και την διανομή των αρμοδιτήτων ως προβλέπονται στον λόγο άρθρο. Εγώ μπήκα και στις αρμο... έμεινα στις αρμοδιότητες επιτροπής μας ε, κάποιες συμπληρωματικές τροπολογίες έχω καταθέσει στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως αφορούν κυρίως ε, διευκρινήσεις και αφορούσαν την προσέγγιση που ακολούθησα στην ε, γνωμοδότηση. Γρήγορα πιστεύω θα μπορέσω να προτείνω τροπολογίες συμβαστικές του συναδέλφους κυρίως για τα άθρα 6, 9 και 10. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, διότι μάλιστα πολλοί συντάκτες των τροπολογιών απουσιάζουν από την αίθουσα σήμερα, άρα θα ήταν δύσκολο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τους παρόντες συναδέλφους και που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Και τους ευχαριστώ και των προτέρων. Okay, Καλώς. Δεν υπάρχουν και πολλοί παρόντες, λέει ο Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα τα πάμε όμως. Κάποιος από τους σοσιαλιστές θέλει να πάρει το λόγο, όχι. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Για τον κύριο Μπουζόη. Ο κ. Μπουζόη ζητά συγγνώμη που απουσιάζει από τη συζήτηση όσον αφορά τις τροπολογίες για την γνωμό της κυρίας Γκαλούρ. Την ευχαριστεί για την επικοδομητική συζήτηση τον οποίο, της οποίας ηγήθηκε πριν υποψήφιων τροπολογίες υπέβαλε κάποιες τροπολογίες δικές του και κάποιες μαζί με τον κύριο Κρόιτσμαν. Κάποιες τροπολογίες αφορούσαν τη νομική αξία των ειδικών αυτών ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων. Πιστεύει ο κ. Μπουζόη ότι είναι παραπλανητικό κάπως στιγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως να δίνει υψηλότερο ε, νομικό καθεστώς όσον αφορά την ηλεκτρονική σφραγίδα από ό,τι δίνει ο Εθνικός Νόμος για τους φυσικές σφραγίδες. Η τροπολογία του κυρίου Μπουζόη το διευκρινίζει αυτό για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση. Άλλη πτυχή, η νομική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων, η αναφορά στο επίπεδο ακεραιότητας και αυθεντικότητα, το εξασφαλισμένο επίπεδο αυθεντικότητα, είναι κάτι που παραπλανεί. Μπορεί να ακολουθεί η ίδια προσέγγιση όπω και για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ, ηλεκτρονικέ φραγίδες και χρονογραμματώσιμα και θα λέει ότι δεν θα πρέπει να, να μην έχουν νομική ισχύ τα έγγραφα τα ηλεκτρονικά επειδή είναι ηλεκτρονικά. Αλλά παρόλα αυτά να αλλάξει διατύπωση θα δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Η νομική συνέπεια των ηλεκτρών εγγράφων που έχουν κάποια ηλεκτρονική υπογραφή εγκεκριμένη ή κάποια εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα η ισχύ του πρέπει να είναι ίδια με ένα φυσικό χαρτί που έχει χειρόγραφη υπογραφή ή φυσική σφραγίδα υπό τη στιγμή που τα έγγραφα δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε ε, αυτομάτως, ούτε διαφορετικά. Υπέβαλε και άλλες ε, τροπολογίες για ελαχιστοποίηση των στοιχείων μαζί με τον κ. Κρότσμαν. Οι υπηρεσίε διαφέρουν τη φύση τους, ποικίλουν και ίσως να χρειάζονται διαφορετικά προσωπικά στοιχεία για ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Γι' αυτό θεωρείται λογικό να απαιτούνται μόνο τα στοιχεία που είναι απόλυτα αναγκαία για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Παραδείγματο χάρη, αν μόνο η ηλικία είναι σχετικό στοιχείο, δεν έχει νόημα να απαιτούνται και άλλα προσωπικά στοιχεία, διότι τα στοιχεία αυτά ούτω ή άλλω δεν είναι χρήσιμα στα πλαίσια συγκεκριμένη υπηρεσία. Και τέλο, εξίσου σημαντικό, και ο Μπουζόη θέλει να κάνει κάποια σχόλια όσον αφορά τι διατάξει που αφορούν του εποπτικού φορεί. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό το όνομα τη εποπτική αρχή, καθώ και τα στοιχεία για επαφέ με του αρμοδίου αυτού του ελεκτικού φορέα θα πρέπει να κοινοποιούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμη πιο σημαντικό δεν θα πρέπει να γίνεται μνήμα στις ερευνητικές εξουσίες διότι αυτές ίσως να αφορούν μόνο τις αρχές επιβολής του νόμου. Τα καθήκοντα των εποπτικών φορέων αναφέρονται σαφώς στον κανονισμό και αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι φορείς αυτοί έχουν τις αναγκαίους πόρους ούτως ώστε να διενεργούν ε, αυτές τις έρευνες, να, ασκούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά την αμοιβαία αρρωγή μεταξύ εποπτικών φορέων οι εποπτικοί φορεί θα πρέπει πράγματι να ανταλλάσσουν βέλτιστε πρακτικέ, αλλά θα πρέπει να ζητούν αμοιβαία αρρωγή μόνο σε δικαιολογημένε περιπτώσει, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα τη ε, εργασία του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κ. Σάγκστρομ. Μερικά σύντομα σχόλια για τα δεδομένα Κοιτάξτε, εγώ βλέπω με πολύ ενδιαφέρον αυτές τις τροπολογίες, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πτυχή στο σχεδιασμό τέτοιου είδους πραγμάτων. Ε, στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων ε, που είχαμε, συζητήσαμε την τιμή. Να ξαναπώ αυτό που είχα πει και τότε. Δεν θέλω να βρεθούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την ταυτοποίηση πρέπει να πληρώνουν γι' αυτό. Με μια αναλογική κάρτα ταυτοποίησης ε, μπορεί να πληρώσει κάποιος ε, για να την ε, λάβει, αλλά μετά δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτε επιπλέον. Αν οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν, αν αλλάζουν χρήματα χέρια, όταν χρησιμοποιείται η κάρτα αυτή, θα μπορούσε να είναι επικερδές κάτι τέτοιο για κάποιους φορείς που μπορεί να προσπαθήσουν να το χρησιμοποιούν αυτό στο δυνατόν περισσότερο και αυτό αντίκειται ε, στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Και στην αρχή αυτή ναι, καλό είναι αυτό να το κάνουμε, ε, αλλά δεν θέλουμε να ε, χρησιμοποιείται κατά κόρον σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε. Και είναι κάτι ακόμη το οποίο με απασχολεί, γι' αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Όμπερμαϊρ. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν Μία πολύ θετική, θα έλεγα, ιδέα σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία. Στις τροπολογίες δηλαδή, να συμπληρώσω απλά και μόνο ότι το ουσιώδες είναι η νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα στην οποία πρέπει να μπορεί να βασίζεται κανείς και για τις ανησυχίες ή επιφυλάξεις που υπάρχουν σε σχέση με τους διάφορους όρους και προϋποθέσεις δεν μπορεί να είναι αρκετά αυστηρά αυτά τα πλαίσια. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να δούμε είναι η δεδομένη αποδοχή αυτών των δυνατοτήτων. Αποδοχή με ηλεκτρονική ταυτότητα ή κωδικό με τον οποίο πρέπει να μπορούμε να εργαζόμαστε για να δοθεί μια απάντηση σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Είναι ένα ωραίο πράγμα στο οποίο μπορεί να αναφέρεται κανείς σε φοιτητέ στα πανεπιστήμια με αποτελέσματα πειραματικά που διασυνοριακά μπορούν να αποστέλλονται από τη μια χώρα στην άλλη. Θετικό είναι αυτό, αλλά δύσκολο είναι να συγκρίνουμε όλα αυτά με ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Αυστρία μια ιδέα ε, ιατρικής κάρτας για παράδειγμα που δεν, δεν χρησιμοποιείται στην Ευρώπη όταν περνά κανείς ως ασθενής από μια χώρα σε άλλη να υπάρχει ένας αριθμός, ένα, ένας κωδικός ο οποίος δεν θα αγνοείται από τους γιατρούς που εργάζονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχει ένας δεσμευτικός χαρακτήρας που θα συνδέεται και με κυρώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε όλες οι χώρες ε, να μπορούν να τα αποδέχονται αυτά και να μπορούν να τα εφαρμόσουν σε σχέση με το πλαίσιο εφαρμογής. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάποια σχόλια μόνο και σε σχέση με την κυρία Γκάλο στο πλαίσιο σκιωδών εισηγητών. Ήμουν πάντα πολύ επιλεκτικό σε σχέση με τις τροπολογίες επικεντρούμενο σε θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι θέματα αρμοδιότητάς μας όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά, κυρίως για το πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν και θα λειτουργήσουν και ποιος θα είναι ο ρόλος των αρμόδιων αρχών για τα επίπεδα, για παράδειγμα, ποια κεντρική εποπτεία είναι, ανάγκη, ώστε να, ε, ε, είναι αναγκαία ώστε να μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν και σε συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών για να κινηθούμε ταχύτερα. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε ως Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά για να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Μου φαίνεται μέρος του προβλήματος είναι ακριβώς εδώ το ότι είχαμε αρχικά μία οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές του 1999. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα στα οποία εργάστηκα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, στο τέλος της θητείας μου ξαναεργαζόμαστε επ' αυτού του θέματος. Δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, τεράστια πρόοδος όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικές φραγίδες με την ενθάρρυνση των χρηστών ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να στεφθούν με επιτυχία στις αγορές. Το πραγματικό θέμα είναι πώς θα κινητοποιήσουμε κινητοποιηθούμε προς τα εμπρός και θα τα προαγάγουμε όλα αυτά για να στεφθούν με επιτυχία. Ποια θα είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν από τα κράτη-μέλη για να υπάρξουν επενδύσεις στις υποδομές για να λειτουργήσουν αυτά σωστά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αναφέρουμε λοιπόν κάποια σημεία τα οποία θίγουμε για τις περίπλοκες πτυχές ε, που ε, συναρτώνται εδώ και για το φιλόδοξο πλαίσιο που σίγουρα θα πρέπει να είναι φιλόδοξο. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε και το πώς θα σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει δέσμευση επ' αυτού και από τους παρόχους και σε σχέση με όσους ε, θα συνεργαστούν για να κινηθούμε με τους δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς. Επ' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο κύριος Κρόιτσμαν έχει καταθέσει αρκετές πολλές τροπολογίες ο ίδιος και νομίζω πορεύονται και στοχεύουν και προς ε, την κατεύθυνση που θα θέλαμε εμείς να κινηθούμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Άλλος που θα ήθελε να σχολιάσει επ' αυτόν, παρακαλώ. Ίσως να ζητήσω τώρα εσάς ε, κύριε Σαβίδη να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις για αυτές τις τροπολογίες και θα επανέλθω στην κυρία Γκάλο και με το χρονοδιάγραμμα. Εσείς κύριε Ιακωβίδη παρακαλώ. to um, the committee. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, τους συζητητές ε, ε, και όλους όσους ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Πράγματι φαίνεται ότι συμφωνούμε στον τρόπο με τον οποίο αυτός, αυτή η νέα νομοθεσία μπορεί να ε, βελτιώσει ε, την εμπιστοσύνη στις ε, ψηφιακές αγορές. Κάποιες από τις τροπολογίες πιστεύουμε ότι θέτουν σημαντικά θέματα σε σχέση με ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως η ασφάλεια δικαίου επειδή είμαστε σε πλαίσιο κανονισμού ευχαρίστως να συνεργαστούμε με, τον με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές ε, για ε, να δούμε ε, πώς είναι δυνατόν αυτές οι συμβιβαστικές τροπολογίες να είναι αποτελεσματικές. Υπάρχουν κάποιες πτυχές βέβαια σε σχέση για παράδειγμα με το ρόλο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που απομακρύνονται κατά τη από, την, από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχει ας πούμε το βασικό επιχείρημα της επαρκούς ε, ασφάλειας και της ε, χρήσης των δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνη και την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πολύ επικοδομητική η δουλειά που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γκαλό. Χαίρομαι που όλος ο κόσμος είναι αισιόδοξο ε, και χαίρομαι επίσης ε, γιατί πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ε, είδαμε πολύ προσοχή της τροπολογίες του συναδέλφου Μπουζόη, ο οποίος δεν θέλει στα ηλεκτρονικά έγγραφα να δώσει μεγαλύτερη σημασία από ότι τα ε, φυσικά έγγραφα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως αυτονόητο βέβαια, ε, αλλά όλες αυτές οι τροπολογίες βεβαίως ε, λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, όσον αφορά την ελαχιστοποίηση των δεδομένων είναι και αυτό μια σημαντική αρχή και θα ήθελα να καθησυχάσω τον συνάδελφο Έγκστρομ και αυτό θα το προσέξουμε και είναι βέβαια μια ανησυχία που μας απασχολεί, που την έχουμε και εμείς. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή και στις δικές σας τροπολογίες για την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι συχνά τροπολογίες ε, που ο συνάδελφος Σφάμπ ε, έχει επίσης υποβάλει. Στο γαλλικό δίκαιο, για παράδειγμα, δεν λέμε ότι πρέπει κανείς να έχει την απόδειξη ότι δεν έχει διαπράξει αμέλεια, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στο πλαίσιο του γαλλικού δικαίου μια αρνητική απόδειξη. Λέμε ότι κάποιος ε, λέμε, λέμε ότι κάποιος ε, πρέπει να επιφέρει μία απόδειξη ε, η οποία να είναι θετική. Εν πάση περιπτώσει ε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Νομίζω δηλαδή ότι θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για το χρονοδιάγραμμα ότι η δική μας εμείς θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο, αλλά η Ήτρε θα ψηφίσει το Σεπτέμβριο. Οπότε, τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και παραμένω και εγώ πολύ αισιόδοξη σε σχέση με το συμβιβασμό. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε ποιες θα είναι οι συμβαστικές σας προτάσεις για τον Ιούλιο και περιμένουμε σαν μέρος Επιτροπής Βιομηχανίας να προωθήσετε... Α, δεν είσαστε, είσαστε. Α, να προωθήσετε τις δραστηριότητε μας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αυτό ήθελα να πω. Θα είναι πολύ σημαντικό. Ορότατα, καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και παρίσταται εδώ σήμερα το απόγευμα. Προχωράμε και πάμε στο τελευταίο σημερινό μας σημείο, δηλαδή πρόταση ψηφίσματος που σχετίζεται με στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ασφαλής και ασφαλής κυβερνοχώρος. Υπενθύμηση. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας για το πακέτο για τις, ε, για τις πληροφορίες και την ασφάλεια και αύριο έχουμε ακρόαση σχετική. Όλοι είστε πρόσδεκτοι να παραστείτε, στις 3 ώρα θα γίνει ακρόαση και σαν ένα τμήμα του πακέτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει ένα, τα, ετοιμάσει ένα γενικό ψήφισμα, μία γίδα, ένα πλαίσιο. Ένα κείμενο μη νομοθετικό που καθορίζει σαφώς μια στρατηγική προσέγγιση για τον απανή, ανοιχτό και ασφαλή κυβερνοχώρο. Συμπεριλαμβάνονται και άλλες πτυχές πλέον της ασφάλειας, πέραν της ασφαλείας. Θέλαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, στο έγγραφο αυτό, υπό τη μορφή ενός ψηφίσματος από πλευράς Κοινοβουλίου, διότι θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια αντίδραση, παράλληλα αυτό με την νομοθετική μας εργασία και υπάρχουν διάφορα ζητήματα που τίθενται. Ο, η κυρία Βερχέιεν θα μας παρουσιάσει ε, εκ μέρους του Άντριου το κείμενο. Θα υπογράψω και εγώ ε, σαν πρόεδρος Επιτροπής το κείμενο. Έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος και τις σχετικές τροπολογίες. Ο κ. Γασίας Φερμόν ε, συμμετέχει από πλευρά σοσιαλιστών, ο κ. Μάντερ, ο κ. Μαρκάκη, θα μιλήσει για τους φιλελευθέρους και ο Κρίστιαν Έγκστρομ και εγώ θα πάρουμε το λόγο και η κυρία Μακλάρκεν που ασχολείται σαν σκιώδης με το θέμα αυτό. Η κυρία Βερχέιεν θα κάνετε εκ μέρους του κυρίου Άντριου Σβάμπ μια παρουσίαση. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του Ανδρέα Σβάβ, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί. Και εκπροσωπώντας τον σύντομα θα πω δύο λόγια για το, την πρόταση ψηφίσματος για την κυβερνοασφάλεια. Υπήρξαν 129 τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους. Συμπεριλαμβάνονται και εκείνες από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές Ήτρε, Λίβε, Ιντερν και από την ΑΦΕΤ εξωτερικών υποθέσεων αναμένονται τροπολογίες για την άμυνα στις κυβερνοεπιθέσεις. Θέλει να ευχαριστήσει για όλες τις τροπολογίες ο συνάδελφος ΣΒΑΜ, ιδιαίτερα και για τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που κατέθεσαν τροπολογίες. Ευχαριστεί για την θετική συνεργασία και τις ενδιαφέρουσες προτάσεις και παρατηρήσεις που γίνονται. Μετά από μια πρώτη ε, μελέτη, περίπου 15-17% ε, αφορούν το θέμα της κυβερνοεγκληματικότητας και έτσι θα έπρεπε να δούμε το κατά πόσον μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο για την κυβερνοεγκληματικότητα και όχι τόσο για την κυβερνοασφάλεια. Η στρατηγική κυβερνοασφάλεια, όμως, όπως αναφέρει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει και άλλες πτυχές τι πτυχές της βιομηχανίας, ε, την διεθνή πολιτική, όλα αυτά πρέπει να ε, βρίσκονται σε μια σωστή ισορροπία λοιπόν. Στις τροπολογίες πολλές καλές προτάσεις εμπεριέχονται που ο Ανδρέας Σουάμπ σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται. Για παράδειγμα τον κέριο ρόλο της ε, ιδιωτικής ε, ε, δημόσιας εταιρικής σχέσης και που από πλευρά στη Ήτρε ή για παράδειγμα αμφίδρομα θα πρέπει να δράσουμε όπως από πλευρά του συναδέλφου Λόπε Θαγγιλά ή και από τους σοσιαλδημοκράτες και από την Λίμπε κατατίθεται ως πρόταση παρόμοια τροπολογία μάλλον και από την ΑΦΕΤ θα κατατεθεί. Σε κάποια σημεία ο Ανδρέας θα ήταν ευγνώμων αν θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν κάποιες επεξηγήσεις, περαιτέρω επεξηγήσεις, για παράδειγμα για την εκφώνηση συμβιβαστικών τροπολογιών. Υπάρχει μια τροπολογία Γκασές Ραμών για παράδειγμα, η τροπολογία 14, η 41 και 99. Στην 99 ιδιαίτερα το θέμα τίθεται αν θα επιθυμούσε τα κράτη-μέλη την σύμβαση της Βουδαπέστης να την κυρώσουν ή όχι. Ή μήπως εννοεί ότι ένα νέο μέσο πρέπει να δημιουργηθεί. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ ο Ανδρέας Σβάπ θα προτιμούσε μάλλον τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν, να κυρώσουν τη σύμβαση της Βουδαπέστης περισσότερο. Κατά τούτο λοιπόν χρειάζονται κάποιες αποσαφηνήσεις, κάποιες διευκρινήσεις και θα τον ικανοποιούσε τον Ανδρέα Σβάμπ αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα και έχουμε και μια τροπολογία την 19 έχουμε του συναδέλφου Άγκστρομ όπου πρόκειται για ένα σύστημα που πρέπει να αντιμετωπίσει failures. Θα ήθελε ο Ανδρέας Σουάπ να γνωρίζει περί τίνος ακριβώς πρόκειται, να μας δοθούν κάποιες επεξηγήσεις. Υποβάλλονται και κάποιες προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες που ε, θέλει να υποβάλει ο Ανδρέας Σουάπ ως εισηγητής. Ο Ανδρέας θα χαιρότανε αν σε μικρή προθεσμία θα ήταν δυνατό να έχει τις προτάσεις σας ώστε το χαρτοφυλάκιο να ολοκληρωθεί και να μπορέσει να υποβάλει τέτοιου είδους συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Γασίας Φερμόν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξίσου και εγώ όπως και ο προλαλή θα ήθελα και εγώ να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόταση ψηφίσματος μεγάλης εμβέλειας, μεγάλης σπουδαιότητας Πράγμα που μας υποχρεώνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να εξετάσουμε σε βάθος ε, τις συνιστώσεις που θα εντάξουμε στις τροπολογίες και προτάσεις που καταθέτουμε και το πώς θα αντιμετωπιστούν. Φυσικά είμαι πρόθυμος να συζητήσω αυτά τα θέματα σε σχέση με την πρόταση που έγινε. Για τροπολογίες δηλαδή που έχω καταθέσει εγώ να δώσω από διευκρινήσεις και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες κάποιων συμβιβασμών, συμβαστικών λύσεων. Φυσικά όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος θα έχει επιπτώσεις και θα αφορά ιδιαίτερες ευαισθησίες και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και πέρα από τις πέντε τροπολογίες που έχω καταθέσει υπάρχουν θέματα σημαντικά που πρέπει να αναζητηθούν. Να αναζητήσουμε ένα ψηφιακό πλαίσιο ασφαλές και βιώσιμο και αξιόπιστο που θα διασφαλίζει και τις ελευθερίες έκφρασης, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων επίσης και τα δικαιώματα στην ιδιωτική σφαίρα, στην ιδιωτική ζωή και την προστασία αυτών των προσωπικών δεδομένων. Χωρίς αυτές τις εγγυήσεις θα καταλήγαμε σε έναν λαβύρινθο πολύ ε, επικίνδυνο. Και γι' αυτό αυτό που θέτω και προτείνω είναι να διευρύνουμε την ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων αυτών, των κιτάρων αυτών στις χώρες όπου δεν υπάρχουν και να ενδυναμώσουμε, να εντείνουμε τις επενδύσεις προς την ανάπτυξη με μεγαλύτερο, μεγαλύτερη καινοτομία. Επίσης τίθεται ότι είναι αναγκαία μια αξιολόγηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών και μέσα σε αυτό το μέτρο να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης μεσοπρόθεσμα που θα εξετάζει προδιαγραφές για την κυβερνοασφάλεια συνολικές και ουδέτερες, αμερόληπτες, ώστε να είναι αξιόπιστες και λειτουργικές. Επίσης, τονίζουμε και την ανάγκη να υπάρξουν κάποιες πολιτικές και ε, στρατηγικής ε, επικοινωνίας ε, για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης ή προειδοποίησης του πληθυσμού. Σε αυτό το μέτρο τονίζω την ανάγκη κατάρτισης και εκπαίδευσης των πολιτών όσον αφορά θέματα κυβερνοασφάλειας. Και ίσως και την ανάγκη του να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης των πολιτών μας προς αυτό το στόχο. Να δημιουργήσουμε και μηχανισμούς εποπτείας και παρακολούθησης. Το, η εγκληματικότητα, το έγκλημα κυβερνοχώρος είναι ένα άλλο στοιχείο και η κυβερνοασφάλεια επίσης. Οι τροπολογίες μου εξετάζουν λοιπόν το πλαίσιο δράσης το οποίο πρέπει να υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να το διατηρήσουμε και σε αυτό το βαθμό οι διαπραγματεύσεις, διατλαντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα και να επιτρέψουν να διασφαλιστούν η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κυριαρχικά της δικαιώματα και αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι προσεγγίσεις και έννοιες, στοιχεία που εμπεριέχονται στις τροπολογίες και φυσικά είμαι πρόθυμος να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα στη συνέχεια και να αναζητήσουμε την ευρύτερη συνένεση. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και ο Σατζημαρκάκης, όχι. Ο Κρίστιαν Έγκστρομ. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 19. Η ασφάλεια χρειάζεται ισορροπία και να καλυφθούν οι κίνδυνοι για να καταρρεύσει το σύστημα. Στις περισσότερες φορές ε, όταν πέφτει το διαδίκτυο δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάτι ποινικό ή επιτίθεται κάποια ξένη χώρα, αλλά γιατί κάτι κατέρευσε, έσπασε. πρέπει να είναι πιο ανθεκτικά τα συστήματα, να μην υπάρχουν σημεία πτώση κατάρρευσης. Καλό αυτό. Και για την καταπολέμηση του εγκλήματο και για την ασφάλεια... αλλά χρησιμότατο για την καθημερινή ζωή. Τα δύο συνδυάζονται. Δεν πρέπει να εστιαζόμαστε πολύ σε πιο περίπλοκους κινδύνους του κυβερνοχώρου και ξεχάσουμε τα απλά πράγματα. Τούτων λεχθέντων. Τροπολογία 120. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή από αυτής. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων το έχουν ρίξει φως στο θέμα αυτό. Ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την περίπτωση κατά την οποία ίσω έχουν διαφορετικά συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ. Τις περισσότερε υποδομές τις ελέγχουν αμερικανικές εταιρείε τι υποδομές μας. Τα συστήματά μα, συστήματα πιστοτικών καρτών κλπ. Κατά πόσο αυτό αποτελεί πρόβλημα. Μετά από τις διαρροές για την NSA και το PRISM και ότι η NSA μαζεύει τόνους ε, πληροφοριών για Ευρωπαίους πολίτες, αυτό δείχνει αυτή την πτυχή. Και πιο συγκεκριμένα, διάβαζα σήμερα κάτι. Σαν τμήμα των επιχειρήσεων του NSA, κατασκοπία κατά των Ευρωπαίων, συνεργάστηκαν με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κλειστών συστημάτων ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν κατονομάζεται εταιρεία. εταιρεία έδωσε πληροφορίες για δυναμίες του λειτουργικού συστήματος στην NSA, ούτω ώστε η NSA να μπορεί να τρυπώσει για κατασκοπία κατά ξένων κυβερνήσεων. Το διάβασα σήμερα αυτό. Εμείς οι Ευρωπαίοι λοιπόν αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Μου αρέσει η Αμερική, δεν λέω. Αλλά πρέπει να είναι φίλοι μας. για να είμαστε σίγουροι ότι παραμένουμε φίλοι, αιωνίως ελπίζουμε, αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να το αξιολογήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Μακλάρκινγκ που είναι η σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μου παρακολούθησε ιδιαίτερα το έγκλημα στον κυβερνοχώρο γιατί είναι μέλος της υποεπιτροπής ε, για το, για έγκλημα σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για τα ε, θέματα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που έχουν να κάνουν με ε, τα παιδιά κλπ. Ε, πολλές αιτιολογικές σκέψεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πρέπει με κοινά μέτρα να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή τόνισε. Όμως υπάρχουμε παγκόσμια, ε, υπάρχει παγκόσμια εγκληματικότητα και παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις, κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε. Το κόστος είναι τεράστιο, στην τροπολογία 2 μάλιστα αναφέρεται αυτό. Ο, το κόστος, το βλέπω στην τροπολογία της, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, 295 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος ε, του εγκλήματος ε, στον κυβερνοχώρο αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο αυτό το ποσό και δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνει, το, αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος πόσο άσχημα είναι τα πράγματα ένα τμήμα του προβλήματος, όπως αναφέρει και στην τροπολογία της 86, είναι ότι σε περικές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές ε, να καταλάβουν ε, την ε, διαφορά ανάμεσα στην νόμιμη και την παράνομη δραστηριότητα, γιατί μερικές φορές και οι παράνομες δραστηριότητες μεταμφιέζονται με πάρα πολύ νόμιμο τρόπο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι και αντικείμενο εθνικής ε, συνεργασίας. Επίσης έχει μία επιπλέον τροπολογία πολύ συγκεκριμένη για, το, για τη Europol γιατί πιστεύει ότι είναι μια επιπλέον, ε, ένας επιπλέον πόρος που μπορεί να μας βοηθήσει με όλο αυτό το πρόβλημα του εγκλήματος στο κυφερνοχώρο. Αυτές είναι λοιπόν οι τροπολογίες της κυρίας Μακλάρκιν. Λοιπόν, θέλει κανένας άλλος να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω τον... τον α, ο κύριος Κάρας και ε, η κυρία Φερχάιεν. Δεν ξέρω εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ή κάποιος. Και μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Φερχάιεν. Έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Χόφερ, εκπροσωπώ την DG Home, μία από τις τρεις μονάδες που εμπλέκονται σε αυτή τη στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια. Ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις με μεγάλη προσοχή τις συζητήσεις και τις τροπολογίες καλωσορίζουμε, είναι καλοδεχούμενες οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες. Γενικά υπάρχει μεγάλη σύγκληση σε σχέση με τα όσα ζητεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τα όσα αρχικά είχε προτείνει η ναι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε τις απόψεις μας αυτές. Θέλουμε να προχωρήσουμε, ε, ο στόχος είναι να προχωρήσουμε παραπέρα λοιπόν στις προτάσεις μας ως εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Home θα ήθελα να καλωσορίσω τις τροπολογίες που αφορούν το κυβερνοέγκλημα αρκετές από αυτές που έχουν κατατεθεί, το γεγονός είναι ότι τονίζουν την ανάγκη να εξοπλιστούμε με τα αναγκαία μέσα και εργαλεία και το επαρκές νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ σοβαρή πρόκληση ή και απειλή κιόλα όπως εκτίθεται. Και φυσικά μπορούμε επίσης ως Γενική Διεύθυνση Home να συμφωνήσουμε με την ανάγκη να υποστηρίξουμε το κέντρο αντιμετώπισης κυβερνοεγκληματικότητας που έχει ήδη εκπονήσει και παράξει αρκετά θετικά αποτελέσματα και είμαστε σε θέση τώρα να αντιμετωπίσουμε υψηλού επίπεδου τέτοιες περιπτώσεις με αρκετά εντυπωσιακά αποτελέσματα σε αυτή την πανευρωπαϊκή ε, δικτύωση για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε να μας δείτε σήμερα το απόγευμα και μας είπατε τις ιδέες σας. Κυρία Περχάιν, θέλετε να ολοκληρώσετε. Να ολοκληρώσω όχι μόνο εκπροσωπώντας κάποιο συμπέρασμα εξ ονόματος του κυρίου Σβάμπα αλλά και προσωπικά θα ήθελα να λάβω τον λόγο και να πω κάτι. Χαίρομαι αφενός για την αποσαφήνιση που δίνεται για αυτή την τροπολογία, για αυτή την χωρίς πρόθεση ας το πω έτσι ε, δυνατότητα να παρισφρέει κάποιο σφάλμα σε αυτό το πακέτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό μέσα στο όλο και μεγαλύτερο έργο ε, που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη δικτύωση. Όλο και περισσότερο στην καθημερινή μας ζωή και στο περιβάλλον μας έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, χειραγώγηση, αντιμετώπιση τέτοιων μηχανών και εξοπλισμών. Πρέπει χωρίς προβλήματα να μπορούν να λειτουργήσουν. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες προδιαγραφές ώστε να υπάρχει αυτή η λειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών και του εξοπλισμού μας στο διαδίκτυο ώστε τέτοιου είδους ε, επιθέσεις εντός εισαγωγικών να μπορούν να αποτρέπονται και να αντιμετωπίζονται ε, στον τομέα ακριβώς δηλαδή της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξησης ε, ε, στο ενεργειακό επίπεδο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναγκαίο να μπορούμε να έχουμε ένα τέλειο συντονισμό. Είναι πολύ σημαντικό για τη σταθερότητα και σταθεροποίηση όχι μόνο των δικτύων αλλά και για όλη την λειτουργικότητα και λειτουργία αυτών των συσκευών και του εξοπλισμού. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και στην εγκληματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε αυτές τις αθέλητες, ας το πω έτσι, σε αυτά τα αθέλητα κενά και προβλήματα που παρουσιάζονται. Είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτό και από πλευρά Έγκστρομ αποσαφηνίζεται επίσης ε, σε σχέση με την ιστορία PRISM και παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων από την NSA στην Αμερική. Θα θέλαμε να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση από τους Αμερικανούς αυτών των θεμάτων και θα χαιρόμαστε αν σε αυτό το σημείο βρίσκαμε λογικές λύσεις που θα οδηγούν οδηγούσαν στο να υπάρξει κάποια εμπιστοσύνη ε, των εταίρων έναντι των Αμερικανών ε, ε, φίλων μας. Αυτά προσωπικά ως παρατηρήσεις. Εξ ονόματος του Ανδρέα Σουβάμπ θέλω να ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις και προτάσεις και για τις πληροφορίες. Νομίζω θα υπάρξει πολύ καλή θετική επικοδομητική συνεργασία για τις συμβαστικές τροπολογίες και θα βρεθούν θετικές λύσεις σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Uh, uh, Θα ήθελα και εγώ να, ευχαριστώ την, να ευχαριστήσω την κυρία Φερχάιεν ε, γιατί μας είπε πολλά πράγματα ε, σήμερα το απόγευμα για το θέμα αυτό. 8 με 9 Ιουλίου θα ε, ψηφίσουμε και θα πάει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες σας τις ιδέες. Δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί το θέμα. Ελπίζω αύριο το απόγευμα να είστε όλοι εδώ, τρει το απόγευμα, όταν θα έχουμε την ακρόασή μας για το θέμα αυτό. Ελπίζω να έρθετε γιατί έτσι θα είναι πιο ενδιαφέρουσα η ακρόαση και πιο ε, πλήρης με τις περισσότερες ε, ερωτήσεις που θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, σημερινή μας συνεργασία, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας ενημερώσατε, ήσασταν και σύντομοι. Να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για σήμερα. Αύριο το πρωί θα αρχίσουμε με την έκθεση της κυρίας Κοράτσα Μπίλ για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Μετά έχουμε από τις 9.45 μέχρι τις 11.15 ψηφοφορία πάνω από, χιλιάδες πάνω από χίλιες τροπολογίες μου λένε ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, πρέπει να ασκήσετε τα δάχτυλά σας σήμερα και αύριο να θυμηθείτε να φέρετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για να μπορείτε να ψηφίσετε. Αύριο 9 η ώρα το πρωί τα λέμε. Γεια σας.